Σας ευχαριστούμε για το σχέδιο γνωμοδότησης που καλύπτει τα πιο βασικά θέματα και ακούσατε και τον υποψήφιο επίτροπο Πίμπαλξ να αναλαμβάνει σχετικές δεσμεύσεις. Λίγα τώρα τεχνικού χαρακτήρα σχετικά με το ΔΕΛΤΑ. Γίνεται αναφορά σε ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ίσως πρέπει να γίνει αναφορά στα εθνικά χρονοδιαγράμματα. Με την έννοια ότι τα εθνικά χρονοδιαγράμματα θα προσφέρουν τους λίθους για να οικοδομήσουμε εμείς το οικοδομημά μας. Τώρα, για τους μηχανισμούς παρακολούθησης στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνούμε απόλυτα με την πρόταση αυτή και συμφωνούμε τόσο πολύ που το κάνουμε ήδη. Ήδη μία φορά το χρόνο την Άνοιξη εκδίδουμε την έκθεση Monterey. για το λεγόμενο monitoring στο συλλογικό επίπεδο. Για το τρίτο εδάφιο τώρα της παραγράφου Α που γίνεται αναφορά σε ενδεχόμενα πρόσθετα προγράμματα Το θέμα που αναφέρεται εδώ, δηλαδή της ε, θνησιμότητας των μητέρων, είναι πολύ σημαντικό. Ίσως όμως η προσθήκη και άλλων μέσων, άλλων εργαλείων για την αντιμετώπιση, ίσως να μην είναι το καλύτερο μέτρο. Ίσως μια ανάλυση ανατομής, και αυτή είναι πολύ σημαντική. Αν όμως προσθέσουμε και άλλους μηχανισμούς, ίσως υπονομεύσουμε την αποτελεσματικότητα των εθνικών μηχανισμών. Κάποια διατύπωση θα μπορούσατε να επιλέξετε χωρίς να προσθέσετε νέους μηχανισμούς. Και νομίζω ότι και οι ειδικοί και οι γιατροί θα το εκτιμήσουν αυτό. Τώρα, συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενωμένων Εθνών. Είναι σημαντικό που εστιάζετε την προσοχή σας στους στόχους της χιλιετίας. Είναι σημαντικό επίσης να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον τομέα της ανάπτυξης, για να επιτευχθούν οι στόχοι της χιλιετίας, γίνεται προσπάθεια από τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά χρειάζεται να υπάρξει μία ενότητα, έγινε κάτι το οποίο ε, το έχει προωθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με θετικά βήματα, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν πρόοδοι και στον τομέα της χρηστής διοίκησης στον τομέα αυτό. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει σίγουρα να, να παίζει ένα ε, ενεργό ρόλο στις εξωτερικές αυτές σχέσεις. Εσείς κύριε Γκερέρο Σαλόμ θέλετε να προσθέσετε κάποιο σχόλιο. Ναι, ευχαριστώ για τις προτάσεις σας και του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Κάποια στιγμή είπα ότι σχεδόν σίγουρα η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ΑΦΕΤ, θα δεχτεί μέρος του δικού μας σχεδίου γνωμοδότησης. Νομίζω λοιπόν ότι το σημαντικό είναι να υιοθετήσει το σημείο Α είναι αλήθεια ότι όσον αφορά τους μηχανισμούς επιπλέον χρηματοδότησης έχουμε αποφανθεί επανειλημμένα εδώ στην Επιτροπή μας με διάφορα έγγραφα. Είναι κάτι που επίσης αποτελεί μέρος μιας γενικότερης, ενός γενικότερου προβληματισμού που έχει να κάνει με την ανάπτυξη και την μεταρρύθμιση των διεθνών χρηματοπιστωτικών μηχανισμών. Άρα θα ενσωματωθεί στην ίδια τη θέση της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ανεξάρτητα με το αν εμείς το ζητήσουμε αυτό ή όχι. Όσο για το τελευταίο σημείο, το σημείο Δέλτα, η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται τόσο πολύ για έκκληση προς τα Ηνωμένα Έθνη, όσο για έκκληση στις ίδιες τις χώρες που αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μέλη πρόκειται για μια δέσμευση που αναλαμβάνουμε προκειμένου να αποτελέσουμε παράδειγμα και να ενισχύσουμε τον ρόλο μας κλειδί στην αναπτυξιακή πολιτική των Ηνωμένων Εθνών. Επιμένω όμως και επαναλαμβάνω, είναι πολύ περισσότερο δέσμευση για τις ίδιες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ίδιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα για την ε, τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκινώ από το τέλος. Η μεταρρύθμιση για την ε, διακυβέρνηση και τα ενωμένα Έθνη πάλι έχει να κάνει με την ε, τοποθέτηση της ΑΦΕΤ. Δεν είναι δηλαδή αναγκαίο εμείς να επιμείνουμε σε αυτό. Να πούμε δηλαδή προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάει η μεταρρύθμιση του Γενικού Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών είναι κάτι που περιλαμβάνεται στην ίδια την θέση και την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της ΑΦΕΤ. Όσο τώρα για την υγεία των γυναικών, των μητέρων, όπως λέει και η Επιτροπή, επικεντρωνόμαστε στο πρόβλημα χωρίς όμως να δίνουμε την ευκαιρία για γενικά προγράμματα που ενισχύουν τους στόχους. Είναι κάθε χώρα χωριστά οι διάφοροι οργανισμοί που φροντίζουν για την τήρηση της δέσμευσης αυτής και την επίτευξη αυτού του στόχου. Πρόεδρος, θυμίζω ότι η κατάθεση για τροπολογίες είναι μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβομημένες χώρες, τροποποίηση του κανονισμού 1934 του 2006. Είναι χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες. Είχαμε ήδη συζήτηση και ψηφοφορία το φθινόπωρο που μας πέρασε, αλλά έρχεται και πάλι αυτή η υπόθεση μπροστά μας επειδή τώρα ισχύει η Λισαβόνα. Χάρη λοιπόν στη νέα συνθήκη, το κοινοβούλιο μας έχει κάτι παραπάνω να πει για το χρηματοδοτικό αυτό μέσο βάσει της νέας νομοθετικής διαδικασίας. Η αλλαγή αυτή έγινε και με νομική βάση που σημαίνει ότι η Επιτροπή μας πρέπει να επανεξετάσει τη θέση της. Το χρηματοδοτικό αυτό μέσο έχει να κάνει με το άρθρο 209 της νέας συνθήκης που μιλάει για την αναπτυξιακή πολιτική. Βάσει όλων αυτών λοιπόν η Επιτροπή μας ζήτησε την εφαρμογή του άρθρου 50 που αρνήθηκε η Επιτροπή Ιντα, που είναι αρμόδια επί της ουσίας. Οι συντονιστές συζήτησαν για αυτό το θέμα και για τη σχετική διαδικασία σήμερα το πρωί και το αποτέλεσμα θα σας το παρουσιάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Σας επικεντρωθούμε λοιπόν τώρα στο περιεχόμενο και δίνω το λόγο στον κύριο Ντέβα που είναι ο εισηγητή μας για πέντε λεφτά. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. η συζήτησή μας για το ε, εργαλείο αυτό θα πρέπει να γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντίθετα με τη συζήτηση που έγινε το 2006, τώρα θα πρέπει να μπούμε και στην ουσία και στην διαδικασία για να ελέγξουμε το, την εφαρμογή του μέσου. Ε, βλέπετε από το κείμενο ότι Πήρα την τελευταία ε, γνωμοδότηση ε, ω σημείο αφετηρία, ω υπόθεση εργασία. Έκανα κάποιε τροπολογίε που προκύπτουν από την αλλαγή τη νομική βάση που προτείνει η Κομισιόν μετά τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα. Συνολικά προτείνω ε, να στείλουμε τρία βασικά μηνύματα. Καταρχά, η Επιτροπή Ανάπτυξη ε, έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την εφαρμογή αυτού του μέσου στι αναπτυσσόμενε χώρε και να χρηματοδοτήσουμε ε, προγράμματα που δεν πληρούν τα κριτήρια της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, ενώ αυτό το μέσο έχει καθαρά, η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια έχει καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα. Το θέμα είναι πώς θα χρηματιδοτήσουμε τα προγράμματα, τις αποστολές που δεν είναι καθαρά αναπτυξιακά. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα 108 εκατομμύρια ευρώ που ε, αρχικά είχαν προβλεφθεί για τη συνεργασία ε, δυνάμει του DCI. Εμείς δεν θέλουμε να δοθούν αυτά τα κονδύλια με αυτόν τον τρόπο. Ε, όπως συμφωνήσαμε πέρυσι όλοι, κάθε ε, ευρώ το χρειαζόμαστε απεγνωσμένα για αναπτυξιακούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να πηγαίνει σε μη αναπτυξιακούς στόχους. Ε, λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι συνολικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υλοποιηθούν και αυτό να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα για τις στοχότερες χώρες. Παράλληλα, οι ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών είναι όλο και μεγαλύτερες. Και φυσικά ε, η πρόοδος στους στόχους της χιλιετίας μπορεί τελικά να μην επιτευχθούν ε, καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν ε, δεσμευόμαστε ότι η γεωγραφική, τα γεωγραφικά ποσά του DCI δεν θα πρέπει να τα αγγίξουμε καθόλου. Το σημείο 2. Η βάση της συνθήκης, όπως είπε και η Κομισιόν, είναι το άρθρο 209 της συνθήκης της Λισαβόνας για τη συνεργασία την αναπτυξιακή. Αυτή είναι η νομική βάση του μέσου. Η νέα συνθήκη δεν αφήνει πολλές εναλλακτικέ λύσεις ε, για μας την Επιτροπή Ανάπτυξη η χρήση αυτού του άρθρου δεν είναι ιδανική λύση, γιατί τα μέτρα που χρηματοδοτεί το ICI δεν πληρούν τα κριτήρια της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Γι' αυτό λοιπόν ε, τονίζω στην αιτιολογική μου έκθεση ότι αυτή η χρήση του άρθρου θα πρέπει να είναι μια εξαιρετική χρήση και όχι συνηθισμένη. Παράλληλα, η συμπερίληψη του 209 ε, έχει οπωσδήποτε συνέπειες. Πρότεινα λοιπόν κάποιες αλλαγές που ξεκαθαρίζουν ότι οι αποστολές στι αντισώμενες χώρες μέσω του, όσο χρηματοδοτούνται μέσω του ICI θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν έναν έμεσο, ε, μια έμεση σχέση με την ανάπτυξη. Η συνέπεια με τις ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τηρηθεί με αυστηρότητα. Τρίτον, δημοκρατικός έλεγχος το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει επαρκή έλεγχο για τον, την εφαρμογή του ICI. Είναι πολύ σημαντικό δεδομένο του αόριστου χαρακτήρα των στόχων και των ε, αποστολών που περιγράφονται. Ε, η διαδικασία που προβλέπεται στο 209 της Συνθήκης Λισαβόνας για τις λεγόμενες εκχωρηθήσεις πράξεις θα πρέπει να αφορά την ε, υιοθέτηση των πολιετών προγραμμάτων υπό το ICI. και η Επιτροπή μας ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ε, για τα πολιετή προγράμματα δυνάμει του DCI. Με αυτή τη δυνατότητα θα ελέγχουμε ε, αυτά τα προγράμματα και θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε σωστά τα χρήματα των φορολογουμένων. Ξέρω ότι η Επιτροπή Ίντα ε, συμμερίζεται αυτή την άποψη και η Επιτροπή ΑΦΕΤ. Δεν έχω υποβάλει συγκεκριμένες τροπολογίες για αυτό το θέμα, αλλά στην επεξηγηματική μου έκθεση τονίζω ότι κάνουμε όσες προσπάθειες μπορούμε για να υπάρξει μεγαλύτερος δημοκρατικός έλεγχος και λογοδοσία. Ευχαριστώ. Το λόγο έχουν οι βουλευτές. Κύριος Μπέρμαν, ευχαριστώ την, τον εισηγητή για την σαφή του παρουσίαση. Όλοι συμφωνούμε με αυτά που είπε ο κύριος Ντίβα. Μόνο μια ερώτηση έχω να θέσω. Είχατε καμία επαφή με τους συναδέλφους ε, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Εμπορίου, ΑΦΕΤ και ΙΝΤΑ, για τη χρηματοδότηση και όλα τα θέματα χρηματοδότησης και την χρήση των κονδυλίων για την ανάπτυξη που πηγαίνουν τελικά σε άλλους στόχους. Πρέπει να έχουμε, και συμφωνούμε σε αυτό, ότι ε, πρέπει να έχουμε ευρία πλειοψηφία ε, στην Ολομέλεια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτές τις επαφές. Προσπαθούμε να κάνουμε λίγο λόμπινγκ, ε, να πιέσουμε τα πράγματα, να πιέσουμε τα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Το έχουμε συζητήσει, όπως ξέρετε, στη συζήτηση των συντονιστών, αλλά η ίντα επιμένει στις θέσεις της. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τους στοχότερους στον αντισόμενο χρόνο. Δεν είμαστε αρκετά δυνατοί για αυτά τα θέματα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ισχύ, γιατί νομίζω ότι έχουμε δίκιο από ηθικής απόψεως. Επομένω, η απάντησή σας είναι συνεχίζονται συζητήσει και εγώ προσπαθώ να κάνω την ψυχραιμία μου. Ε, η Κομισιόν επιθυμεί να κάνει σχόλια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν δεν έχει ιδιαίτερα σχόλια. Το πρόβλημα της ε, πηγής χρηματοδότησης, της χρηματοδότησης είναι ένα πρόβλημα το οποίο το είχαμε συναντήσει από την αρχή. Παραμένει. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πραγματικές δυσκολίες για τη χρηματοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων. Όμως η θέση της Κομισιόν, όπως ε, παρουσιάζεται στην πρότασή της είναι ότι παρότι συμφωνούμε για το στόχο και νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά, τουλάχιστον εγώ έτσι καταλαβαίνω, ότι υπάρχει συνένεση ότι πρέπει να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις δραστηριότητες, παρόλα αυτά πρέπει να, δούμε μια, να βρούμε μια λύση για την πηγή χρηματοδότησης. Προς το παρόν δεν είμαστε ε, σύμφωνοι για την πηγή χρηματοδότησης. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα χρήματα του DCI, για ένα τμήμα της πρότασης του ICI συν, αλλά γνωρίζετε την κατάσταση του τίτλου 4. Το 2010 δεν υπάρχει πια περιθώριο. Το 2011, 2012 και 2013 το περιθώριο είναι ελάχιστα, ελαχιστότατο, μικρό. Επομένως πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να βρεθεί μια λύση. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά να μην ξεχνάμε το στόχο. Και θα πρέπει να συνεργαστούμε ούτως ώστε να βρούμε μια ικανοποιητική για όλους λύση. Και να σας πω και κάτι ενημερωτικό, το, στο Συμβούλιο τα περισσότερα κράτη-μέλη εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην χρησιμοποίηση πόρων από τον DCI. Παρότι και εδώ έλεγε η πρόταση της Κομισιόν ότι ένα μεγάλο τμήμα αυτών των κονδυλίων που λέγαμε να χρησιμοποιήσουμε προβλεπόταν στο συνολικό ποσό του DCI και απλώς θέλαμε να τακτοποιήσουμε λίγο τα πράγματα από νομική άποψης ε, δεδομένων των αυστηρών κριτηρίων για την χρησιμοποίηση των πόρων του DCI. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα μπορούσε να μας βοηθήσει, αν μας λέγατε έτσι πολύ σύντομα, πώς θα χρηματοδοτηθεί το ICI SIN, Plus. Έτσι, μια ιδέα δώστε μας. Και πού θα πάει. Θα πάει σε εκπαιδευτικά προγράμματα, υποτροφίες σε αναπτυσσόμενες χώρες. Πού θα ξοδευτούν αυτά τα κονδύλια τελικά. Ο κύριος Κασμάρεκ. Συμφωνούμε με τον κύριο Ντέβα. Αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να προκύψουν από τον προπολογισμό της ανάπτυξης. Γιατί αν κάναμε κάτι τέτοιο θα αλλάζαμε εντελώ τη δομή του προπολογισμού. Δεν έχουν καμία σχέση με την ανάπτυξη. Επομένως, συμφωνούμε μετά όσο είπε ο κ. Ντέβα. Κομισιόν για να απαντήσει στον κύριο Ντέβα. Ευχαριστώ. Στην ε, νομοθετική της πρόταση, η Κομισιόν, στο νομοθετικό χρηματοδοτικό δελτίο, αναφέρει λεπτομερώς τους ε, βασικούς στόχους χρηματοδότησης, που είναι ε, τρεις. Καταρχάς, η συνέχιση των ε, προπαρασκευαστικών δράσεων που δημιουργήθηκαν από το Κοινοβούλιο το 2007-2008. Αυτές οι δράσεις χρηματοδοτούνται από το περιθώριο που έχουμε και η Κομισιόν προτείνει να συνεχίσουμε και μάλιστα να επεκτείνουμε αυτές τις προπαρασκευαστικές δράσεις με μια χρηματοδότηση από το απόθεμα, από το περιθώριο που έχουμε. Σε ό,τι αφορά την, ε, α, το Erasmus Mundus, προτείνουμε να δώσουμε χρήματα που προβλεπόταν από τον DCI για το Erasmus Mundus. Εκεί είχατε αντίρρηση. Ε, με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ως επίσημη βοήθεια, δημόσια βοήθεια ανάπτυξης, μιλάμε για όντως για υποτροφίες, για το τμήμα EU Mobility. Το πρόγραμμα Erasmus Mundus είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγών. Όταν οι φοιτητέ λοιπόν ξένοι έρχονται στην Ευρώπη, τα ειδικά Κινέζικα Πανεπιστήμια ζητάνε κάποιοι Ευρωπαίοι φοιτητέ να πάνε στα δικά ε, εκεί. Και στο τρίτο τμήμα που είναι τα υψηλά σχέδια, όπου η Κομισιόν θεωρεί ότι κάποια τμήματα να μην είναι ODA eligible, δηλαδή να μην είναι επιλέξιμα με βάση την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, παραδείγματο χάρη στην Αφρική για την ενεργειακή ασφάλεια ή κάποια προγράμματα ε, για public diplomacy, δημόσια για διπλωματία, που μπορεί να μην πληρούν πάλι τα κριτήρια της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Στο κανονισμό άλλα, ε, πριν το 2007, ήδη χρηματοδοτούσαμε τέτοιες δραστηριότητε, αλλά δεν έχουμε αυτό το κριτήριο το νομικό κριτήριο επιλεξιμότητας της δημόσιας βοήθειας για την ανάπτυξη, της δημόσιας χρηματοδότησης για την ανάπτυξη. Το 2007, 2008, 2009 αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα, όπου τα προγράμματα αυτά με την αυστηρή έννοια δεν είναι πλέον επιλέξιμα. Η Κομισιόν λοιπόν στο αρχικό ποσό, στο ποσό αναφορά, είχε προτείνει λοιπόν ε, αυτό το πράγμα για να συνεχιστούν αυτά τα προγράμματα που ήδη χρηματοδοτούνταν από το 2007. Επίσης δώσαμε και ένα non-paper, έναν επίσημο έγγραφο τον Νοέμβριο στην ε, Επιτροπή. Το έχει λάβει και η Επιτροπή σας φαντάζομαι. Για τους, ε, τις αδρές γραμμές, ε, τους αδρούς στόχους που έχουμε που θέλουμε να υλοποιήσουμε με αυτά τα 176 εκατομμύρια ανά περιοχή. Και πάλι αυτά τα χρήματα παραμένουν ε, στις περιφέρειες. Με την ε, δημονασιονομική κατάταξη ε, λέμε Λατινική Αμερική, Ασία, Κεντρική Ασία. Ε, δεν θα πάρουμε αυτά τα χρήματα αν τα βάλουμε σε άλλο κεφάλαιο του προπολογισμού. Δηλαδή αυτά τα χρήματα παραμένουν σε αυτές τις περιοχές. Για την α, ανακατανομή των κονδυλίων του DCI προσπαθούμε να, να επιλύσουμε το πρόβλημα επιλεξιμότητας ε, του ΝΤΑΚ. Τα χρήματα όμως παραμένουν σε αυτές τις περιοχές. Ο κύριος Ντέβα για μία μικρή παρατήρηση. Ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πλήρη απάντηση. Τι εννοεί ο εκπρόσωπός της όταν λέει πρωτοβουλίες διπλωματικές υψηλού προφίλ. Τι ακριβώς εννοεί. Α, εσείς κύριε Μπέρμαν πρώτα. Ερώτηση. Εδώ και 1,5-2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχαμε πει ανταλλαγέ σπουδαστών είναι πάρα πολύ σημαντικέ στα πλαίσια του Εράσμου Mundus. Ουδή το αμφισβητεί αυτό. Ούτε μπορεί να περιοριστεί μονάχα στην ε, πρωτογενή εκπαίδευση, στην ε, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συγγνώμη. Αλλά δεν πρόκειται για χρηματοδότηση τη αποστολή σπουδαστών δικών μας προ τι αναπτυσσόμενες χώρες με χρήματα από την ανάπτυξη. Αυτό για μας είναι απαράδεκτο. Αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπατε, υπάρχει κάποια τέτοια ε, σκέψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κομισιόν μετά όμως θα περάσουμε αμέσως στο επόμενο θέμα. Τώρα να ε, κατηγορείτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, ότι δημιουργεί χρέη. Α, σας πειράζω, σας πειράζω. Ε, καλά, ευχαριστώ, ναι. Η Κομισιόν έκανε μια πρόταση. Πήρε μια απόφαση που υπενθυμίζω ότι ήταν δύσκολο να λυθεί και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά σε μια ρεαλιστική δημοσιονομική προσέγγιση. Η κατάσταση του κεφαλαίου 4 είναι δύσκολη, όπως είπα και πριν. Πήραμε λοιπόν την απόφαση αυτή. Τώρα για την χρέωση πρέπει να ψάξουμε να βρούμε μαζί μια λύση από πού θα προκύψουν τα χρήματα δηλαδή, από ποια πηγή θα αντλήσουμε τη χρηματοδότηση. Η Κομισιόν βεβαίω είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί και με το Συμβούλιο και μετά με το Κοινοβούλιο. Με στόχο να βρει μια λύση στο πρόβλημα αυτό. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να βρούμε ε, λύση αν υπάρχει θέληση από όλες πλευρές. Ε, αν συμφωνούμε δηλαδή στον αντικειμενικό σκοπό. Και σε ό,τι αφορά τώρα τις διπλωματικές πρωτοβουλίες εννοώ ε, διάλογο, διασκέψεις με τις ε, χώρες αυτές για ορισμένα θέματα. Όπως είπα, διασκέψεις, για παράδειγμα για το Ιράν ή το Ιράκ και επίσης ε, έργα που θα αυξήσουν την ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, στις χώρες αυτές με σχετικά χαμηλή χρηματοδότηση. Για να καταθέσετε τροπολογίες για την έκθεση του κ. Ντέβα έχετε προθεσμία μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου το μεσημέρι και τώρα οι αποφάσεις των συντονιστών που λήφθηκαν σήμερα το πρωί. Στα αγγλικά θα τα πω αυτά. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε ακόμα μια έκθεση πρωτοβουλίας για τα συστήματα υγείας στην Αφρική από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και τώρα με αυτή την πρόταση κλείνει μέχρι νεοτέρας η λίστα των ε, εκθέσεων πρωτοβουλίας. Γνωμοδοτήσεις για τον προϋπολογισμό 2011 πάλι ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες που θα ορίσουν τον ε, εισηγητή Ζητήθηκε επίσης το άρθρο, εφαρμογή του άρθρου 50 με την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχουμε με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για τις εφαρμογές του μηχανισμού ICI και εισηγητή για γνωμοδότηση για την λειτουργία της EEAS. Η αρμόδια επιστουσίας επιτροπή είναι η Επιτροπή Εξωτερικών και εμείς έχουμε ζητήσει να εφαρμοστεί το άρθρο 50. Τώρα, αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας, μετά από την απόφαση για τις ποσοστώσεις. Επανεπιβεβαιώσαμε τις τρεις προβλεπόμενες αντιπροσωπείες με αύξηση αριθμού των μελών από 3 σε 4 που αυτά τα μέλη θα επιλεγούν σύμφωνα με το σύστημα The Hunt. Και ζητούμε έγκριση για μία ακόμη αντιπροσωπεία τέτραμελή για την IT με τους στόχους που καθόρισε ο ε, διαρκής συγητής αναλόγως με τις ε, δυνατότητες. Και αυτά θα τα συζητήσουμε και με την αντιπροσωπεία ε, σχέσεων με την Βουλή της για να, δουν, για να δουν θέματα ανοικοδόμησης της χώρας αυτής. Και σε ό,τι αφορά τώρα τις χρονοθυρίες, τα σλότ, η συντονιστές και η γραμματεία λαμβάνουν τακτικά προτάσεις και από εξωτερικές οργανώσεις για να λάβουν χρόνο στην Επιτροπή μας. Όμως ο χρόνος μας μέσα στο έτος είναι περιορισμένος και βεβαίως πρέπει να διατεθεί για την συνήθη κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Η ανταλλαγή απόψεων με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακροάσεις κλπ. Επομένως εξωτερικές οργανώσεις που έρχονται σε επαφή με μέλη ή με τη γραμματεία για να ζητήσουν χρόνο ε, για την ημερήσια διαταξή μας θα πρέπει ενδεχομένως να προσκαλούνται σε μελλοντικέ ακροάσεις. Αυτά θα αποσταλούν στις οργανώσεις αυτές για να γνωρίζουν ότι η Επιτροπή μας ενδέχεται να τις προσκαλέσει, τις οργανώσεις αυτές, εφόσον ανακύψει κάποιο θέμα σχετικό στο μέλλον. Επίσης έκκληση προς το G20 για μεγαλύτερη δημοσιονομική διαφάνεια. Και συμφωνήσαμε ότι θα αποστείλουμε επιστολή στον Πρωθυπουργό του Καναδά στο όνομα της Επιτροπής Ανάπτυξης στην προπαρασκευαστική φάση της διάσκεψης κορυφής του Τορόντο. Ζητήσαμε να συνδεθεί η Επιτροπή μας με μια δημόσια ακρόαση δηλαδή μαζί με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις 18 Μαρτίου και συμφωνήσαμε γι' αυτό. Θα εκπροσωπηθούμε επίσης στην, AD, στην ομάδα εργασίας AD Asher με ένα τακτικό μέλος και ένα αναπληρωματικό που να παρακολουθήσει τις εργασίες της ομάδας αυτής εργασίας και βεβαίως να αναφέρει μετά τα αποτελέσματα, τα πορίσματα στην Επιτροπή μας. Με γραπτή διαδικασία να ζητήσουμε δηλαδή ε, να εκδώσουμε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και αυτά να αποφασιστούν στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών. Σε ό,τι αφορά την ακρόαση για την Παλαιστίνη, ο κύριος Μπλέερ δέχτηκε να συμμετάσχει ωστόσο μπορεί μόνο το απόγευμα της 22ης Μαρτίου. Άρα θα οργανώσουμε έκτακτη ακρόαση του κ. Μπλε στις 22 Μαρτίου. Και δωρεάν κιόλας. Επίσης οι συντονιστές απεφάσισαν να στείλουν ένα τακτικό μέλος και ένα αναπληρωματικό μέλος στην, στον διατρατικό δια, νομοθετικό διάλογο. Μας μένουν λίγα λεπτά. Το αποτέλεσμα της συνάντησης συντονιστών της 14ης Δεκεμβρίου. Δεν το έχουμε ανακοινώσει αυτό. Θα αρχίσω λοιπόν. Θα αρχίσω και όταν έρθει ο Ισπανός Υπουργός θα διακόψω. Είχαμε λοιπόν έκθεση Α, εδώ τα λέει στα γαλλικά. Ή όχι. Α, νομίζω ότι ε, λέει evaluation, δηλαδή αγγλικά. Α, είναι ένα μείγμα. Για τη συνένεση στο ανθρωπιστικό επίπεδο και στα σχέδια δράση είχαμε αποφασίσει να κάνουμε έκθεση πρωτοβουλία για δύο θέματα. Από το ΕΛΚ, κυρία Στίφλερ, και να εκκινήσουμε την διαδικασία, μόλις αυτό θα καταστεί δυνατό, για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα έκος για την ε, ενδιάμεση αναθεώρηση. Για το 2009, για την κοινοβουλευτική συνέλευση, όπου θα υπάρξει έκθεση πρωτοβουλίας της Προέδρου και συμφωνήσαμε ότι η ομάδα η οποία θα αναλάβει την έκθεση θα διορίσει εισηγητή και που αυτός θα πρέπει να είναι και μέλος της, κοινής, ε, της ε, ε μεικτής κοινοβουλευτικής συνέλευσης για την προσωρινή ε, επανεξέταση των στόχων της χιλιοτίας για το Σεπτέμβριο του 2010 με έκθεση πρωτοβουλίας που θα δοθεί για δύο, έναντι δύο βαθμών στους σοσιαλιστές και δημοκράτες το ίδιο για ε, το πλατό των Ιμαλαίων και του Ιντουκούς και, την, και τις επιπτώσεις από τα διοξίδια του άνθρακος. Πάλι εδώ έκθεση πρωτοβουλίας που λαμβάνει η ομάδα ECR ε, έναντι δύο βαθμών. Για πόλη για το Λαϊκό Κόμμα για τις αντιπροσωπείες στην ε, Ζιμπάμπουε και τη Σομαλία. Σύσταση προς το Συμβούλιο για τις Προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 65η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Γνωμοδότηση με... για την σύσταση της ΑΦΕΤ. Νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν. Επίσης εδώ γνωμοδότηση. Ένας βαθμός. άλδε. Ανθρώπινα δικαιώματα ε, τα, στάντα τα στάνταρ τα οποία θα περιλαμβάνονται στις διεθνείς συμφωνίες, οι εξωτερικές διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής, η προώθηση της απασχόλησης, η ευθύνη των εταιριών, γνωμοδότηση της ενωτική αριστεράς, το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής μετά το 2013, είπαμε εδώ όχι γνωμοδότηση, Για το Resettlement Program, program επίσης όχι γνωμοδότηση. Νομική γνωμοδότηση τώρα με προθεσμία για την έκδοση της νομικής γνωμοδότησης για τα άρθρα 290 και 291 τη FIU για τις οριζόντιες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διαπραγματεύσεις με άλλα θεσμικά όργανα για την εφαρμογή αυτών των ε, άρθρων. Όλα αυτά, λέει η Έχουμε και μια ομάδα συντονισμού εκλογών που διορίστηκε για το 2010 για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και τα συνδικάτα τα είπαμε. Αυτά ήταν. Θα περιμένουμε λίγο τώρα το, πριν αρχίσουμε το επόμενο θέμα, δηλαδή τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας.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 Με μεγάλη ικανοποίηση υποδεχόμαστε εδώ τον Μιγγέλ Μορατίνος, υπεύθυνο για θέματα συνεργασίας και ανάπτυξης της Ισπανικής Προεδρίας. Θα μας μιλήσει λοιπόν για το θέμα αυτό. Αφού το άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας, και τον καθορισμό του μόνιμου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ισπανική Προεδρία θα θέσει τα πρώτα λιθαράκια στη νέα πολιτική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων και της ε, αναπτυξιακής βοήθειας θα υπάρξουν πολυάριθμες προκλήσεις να ε, υλοποιήσουμε για την υλοποίηση της ε, υπηρεσίας εξωτερικών υποθέσεων, την αναπτυξιακή βοήθεια, την αύξηση της βοήθειας των πολιτών μας. Ε, τους έξι επόμενους μήνες ε, της Προεδρίας σας, η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, θα συνεργαστεί στενά μαζί σας για να βρει τις κατάλληλες απαντήσει απαντήσεις στις διάφορες αυτές προκλήσεις. Και να πω και ένα τελευταίο προσωπικό σχόλιο. Είχα την ευτυχία να δουλέψω με τον Ισπανό Υπουργό Ανάπτυξης για ένα θέμα που όλοι γνωρίζουν ότι με ενδιαφέρει τα μάλα, τους φορολογικούς παραδείσους και είμαστε απόλυτα στο ίδιο μήκο κύματο ε, ως προς τις απόψεις μας για αυτό το θέμα. Κύριε Μορατίνος, έχετε το λόγο για 20 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, δεν θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ στη δικιά σα Επιτροπή. Σήμερα το πρωί ξεκίνησα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και είπα ότι η παρουσία μου εδώ λαμβάνει η χώρα εκτάκτος, γιατί βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο περιμένοντας την παρουσίαση της έκθεσης της ΥΠΑ του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Είναι απόφαση που θα λάβει το Συμβούλιο για αυτή την ε, Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Λοιπόν, μιλάμε για την ανάπτυξη. Είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο στον ε, προγραμματισμό και στην εκτέλεση της πολιτικής μας αυτή η δικιά σας κοινοβουλευτική επιτροπή. Αλλά όλα αυτά θα φανούν καλύτερα όταν έχουμε την έκθεση της ΥΠΑ του εκπροσώπου. Κυρίε και κύριοι, θέλω να ξεκινήσω την παρουσίασή μου λέγοντα ότι ο αγώνα για την καταπολέμηση τη φτώχεια είναι μια απόλυτη προτεραιότητα στο πρόγραμμα τη Ισπανική κυβέρνηση ήδη από το 2004. Και αυτό θα συνεχιστεί βέβαια και στην Προεδρία μα επιβεβαιώνει και τις προσπάθειες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα άνευ προηγουμένου και αντικατοπτρίζεται και στις αλλαγές που έχουν γίνει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά από πλευρά τη Ισπανία στα θέματα συνεργασίας και ανάπτυξης. Και θέλουμε να μπορούμε να στηριχτούμε και στη δικιά σας Επιτροπή. Κάποιες από τις προτεραιότητες μας έχουν εμπνευστεί από τη δουλειά και τον προγνωστικό ρόλο που έχουν παίξει τα δικά σας ε, τα μέλη και η Πρόεδρος η κυρία Ζολή σε θέματα κινητοποίησης εσωτερικών πόρων για την ανάπτυξη μέσω του αγώνα κατά της φοροδιαφυγής και των ε, φορολογικών παραδείσων. Κυρίες και κύριοι, όπως είπα ήδη, έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία προεδρία του Συμβουλίου που είχε η Ισπανία μέχρι σήμερα. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές ποιοτικέ και ποσοτικέ στην πολιτική μας ανάπτυξης και συνεργασίας. Η κυβέρνηση της Ισπανίας έχει κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες και έτσι έχει περάσει από την αναπτυξιακή βοήθεια που ήταν το 0,24% του ΑΕΠ το 2004 στο 0,45% το 2008. Ε, μόνο φέτος αυξήθηκε κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ η αρρωγή μας αυτή. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν το καλύτερο στην Ευρωπαϊκή, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και το καλύτερο που είχαμε ποτέ στην Ισπανία. Οι αλλαγέ αυτέ μα έκαναν να είμαστε ένα από του κύριου δωρητέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισπανία σήμερα κατέχει την τέταρτη θέση μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον όγκο τη βοήθεια και την όγδη όσον αφορά το ποσοστό του ΕΠ που δίνει για τη βοήθεια αυτή. Συνεπώ, έχουμε δεσμευτεί προ αυτή την κατεύθυνση και θα συνεχίσουμε. Και παρά την οικονομική κρίση, το επαναλαμβάνω, και παρά την οικονομική κρίση θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο 0,51% του ΕΠ για την αναπτυξιακή βοήθεια το 2010. Έτσι θα τηρήσουμε τον στόχο που είχε θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2005 και θα δώσουμε ένα βήμα παραπάνω για να φτάσουμε στο στόχο του 0,7%. Η συνεργασία για την ανάπτυξη έχει αποτελέσει ένα κεντρικό στοιχείο στην εξωτερική δράση της Ισπανίας και αποτελεί μία πολιτική αυτή καθεαυτή. Έτσι λοιπόν εμείς την Προεδρία αυτή την αναλαμβάνουμε από μια θέση πολύ πιο στέρεα και με πολύ περισσότερες φιλοδοξίες. Θέλουμε κυρίες και κύριοι να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι κατά το παρελθόν και να συνεισφέρουμε στην παγίωση μιας πραγματικής αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρώπης. Θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και συνεπείς με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ισπανία και οι άλλες χώρες μέλη. Όμως αναλαμβάνουμε την Προεδρία αυτή και μέσα σε ένα πλαίσιο πολύ πιο δύσκολο που χαρακτηρίζεται από διάφορου αποφασιστικού τομεί. Πρώτα απ' όλα άρχισαν να ισχύει η συνθήκη τη Λισαβόνα και δεύτερον έχουμε την οικονομική και δημοσιονομική κρίση με τι συνέπειέ τη. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν φτιάχτηκε και το δικό μας πρόγραμμα για το εξάμεινο αυτό, το οποίο όπως καταλαβαίνετε χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία αυτά. Η συνθήκη της Λισαβόνας, κυρίες και κύριοι, σημαίνει αλλαγέ στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, στη διαδικασία οικοδόμησης. Κάτι το οποίο πάντα ήθελε η Ισπανία, πεπισμένη για την ευρωπαϊκή μα διάσταση. Εμεί είμαστε πεπισμένοι ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα αποτελεί στοιχείο κλειδί για μια αναπτυξιακή πολιτική η οποία θα προσανατολίζεται για να καταπολεμήσει την ένδια και που θα βρίσκεται μέσα στο κέντρο των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 21.2. Και η συνθήκη επίσης ενισχύει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ε, κέριο παράγοντα προκειμένου να έχουμε συνεπή πολιτική με τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή σε θέματα συνεργασίας. Η συνέπεια αυτή θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε όλο το δυναμικό που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να είμαστε ο πρώτος δωρητής παγκοσμίω. Συνεπώς, είναι η Ισπανική Προεδρία και η Ισπανία να συνοδεύσει τα πρώτα βήματα της διαδικασίας αλλαγών της θεσμικής αρχιτεκτονικής και της συνεργασίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να φτιάξουμε ένα σενάριο μετά τη Λισαβόνα. Οι αλλαγέ αυτέ θα μα επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα τι δυνατότητε που μα δίνει η συνθήκη. Θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, ενωμένοι και αυτό να φανεί στη δράση μα που να είναι συνεπή απέναντι στου φιλόδοξου στόχου ανάπτυξη που έχουμε. Ω Προεδρία βέβαια αντιμετωπίσαμε την πρόκληση της τεράστιας ανθρωπιστικής καταστροφής στην ΑΙΤΗ. Ήταν η πρώτη πρόκληση που είχαμε τώρα που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε όσο γίνεται καλύτερα τις νέες διατάξεις, τις θεσμικές που περιλαμβάνει η νέα συνθήκη. Δεν υπάρχουν πολλά προηγούμενα όπως αυτή η καταστροφή, τα Ηνωμένα Έθνη μίλησαν για τη χειρότερη φυσική καταστροφή την οποία είχε να αντιμετωπίσει ποτέ σε ολόκληρη την ιστορία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Μπροστά στην κατάσταση αυτή λοιπόν εμείς δουλέψαμε για να καταφέρουμε να έχουμε μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ύψος των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει υπέρ της αλληλεγγύης. Μεγάλη αξία αυτή, βασική αξία μέσα στην ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και έτσι θελήσαμε ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πολύ βασικός ω δωρητή. Από τη στιγμή που πήραμε τα πρώτα νέα για το σεισμό στην Αιτή, η Ισπανική Προεδρία ανέπτυξε όλε τι δυνάμει δυνάμεις για να μπορέσει να συντονίσει και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή δράση. Οι καταστάσει βέβαια ήταν πολύ δύσκολε που αντιμετωπίσαμε και γι' αυτό δυσκολευτήκαμε, αλλά μπορέσαμε να αντιδράσουμε γρήγορα και συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα. Η Γενική Γραμματεία για τη Λατινική Αμερική, η Γενική Γραμματεία για τη Συνεργασία και την Προεδρία τη ε, κυβέρνηση τη Ισπανία, πήγανε στην Ισπανία για να συντονίσουν τη δράση μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την Υπηρεσία για την Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξεκίνησε έτσι μία μονάδα συντονισμού και κατεπίγουσας βοήθειας με πυρογνώμονες σε θέματα όπως αυτό που είχαμε στην ΑΕΤ. Και επίσης φροντίσαμε να υπάρξει και ενίσχυση λογιστική στη διάθεση της ΥΠΑ του εκπροσώπου, της Επιτροπής και των ε, χωρών μελών. Κυρίε και κύριοι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάναμε και θα επανέλθω απαντώντας ερωτήσεις σας δίχως άλλο όταν μιλήσουμε για τον ρόλο που παίζει η εκπεριτροπής Προεδρία και που έπαιξε τις πρώτες στιγμές της τραγωδίας στην ΑΕΤ. Εφ' εξής, κυρίες και κύριοι, πρέπει να είμαστε σε θέση να δρούμε συντονισμένα στην ΑΕΤ, να διασφαλίσουμε την μετάβαση ανάμεσα σε αυτήν τη φάση κατεπίγουσα βοήθεια και τη φάση ανοικοδόμηση τη χώρα. Η Ισπανική Προεδρία προτείνει να δουλέψει όσο γίνεται περισσότερο προκειμένου να πετύχουμε αυτό το στόχο. Κυρίε και κύριοι, όπω είπα και πριν, ο δεύτερο παράγοντα που καθορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται η δικιά μα Προεδρία είναι εκείνο τη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Συνειδητοποιούμε τι έκτακτε δυσκολίε που δημιουργεί η κρίση στι αναπτυσσόμενε οικονομίε οι προβλέψεις που έχουμε από τον ΟΕ στην έκθεση του 2009 για τους στόχους ε, της χιλιετίας υπογραμμίζεται ότι η κρίση και καθυστερεί το ρυθμό προόδου προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, αλλά επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις έχουμε και προς τα πίσω πορεία στόχων οι οποίοι νομίζαμε ότι είχαν πετύχει η πεποίθηση ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η οικονομική κρίση να, δημιουργήσει μια κρίση ανάπτυξης είναι αυτό που προέχει για να καθοριστούν οι προτεραιότητες τη δικιά μα ισπανική προεδρία. Πρέπει να διπλασιάσουμε τι προσπάθειές μα για να πετύχουμε του στόχου τη χιλιετίας. Αυτό απαιτεί στα σημερινά πλαίσια κινητοποίηση όλων των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μα. Να προχωρήσουμε και να τηρήσουμε τι δεσμεύσει του Μοντερέ και τη Δόχα και να αποφύγουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας να χαθούν μέσω φοροδιαφυγής, για παράδειγμα. Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις και του Παρισιού και της Άκρα. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε ε, βάσει των όσων ξεκίνησε η προηγούμενη Προεδρία. Να παγιώσουμε τα κεκτημένα και μαζί με το Βέλγιο και την Ουγγαρία η Ισπανία να θέσει σαν κύριο στόχο τις κατάλληλες απαντήσεις που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις από την κρίση. Κυρίες και κύριοι, οι στόχοι της χιλιετίας, όπως είπα, αποτελούν έναν από τους τρεις άξονες που θα διαρθρώσουν τη δράση μας απέναντι στην κρίση σε θέματα ανάπτυξης. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να δούμε η Ειδική Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για την ε, αναθεώρηση των στόχων της χιλιετίας το Σεπτέμβριο φέτος πού θα καταλήξει προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμευτεί για την επίτευξη όλων των στόχων που η διεθνής κοινότητα έθεσε πριν από ένα χρόνια. Η, Ισπανία θα οθήσει τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της διάσκεψης αυτής του Σεπτεμβρίου σε θέματα ανάπτυξης. Επιπλέον θέλουμε να ετοιμάσουμε μια συζήτηση, πρώτη συζήτηση κυρίες και κύριοι, για πρώτη φορά οι ηγέτες κατών και κυβερνήσεων στο Συμβούλιο του Ιουνίου θα συζητήσουν για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και θα συμπεριλάβουν και τους στόχους της χιλιετίας και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί υπέρ της ανάπτυξης. Έτσι θα τηρηθεί αυτό το οποίο συμφώνησε το Δεκέμβριο που μας πέρασε το Συμβούλιο. Ο κόσμος περιμένει από την Ευρώπη ένα ισχυρό μήνυμα, περιμένει να δεσμευτεί Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη για να πετύχουμε συγκεκριμένες δράσεις στον πρώτο στόχο της χιλιετίας. Δηλαδή, να εκπονήσουμε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική ε, ασφάλειας για τα τρόφιμα. Όπως ε, το γνωρίζετε, η Ισπανική κυβέρνηση σε αυτό το θέμα δίνει προτεραιότητα και έτσι και οργάνωσε και την συνάντηση υψηλού επίπεδου όσον αφορά την διατροφική ασφάλεια στις αρχές του 2009 με ε, πολλά χρήματα για το σκοπό αυτό. Έπειτα όσον αφορά την υγεία και εδώ θέλουμε να υπογραμμίσουμε τη χρηματοδότηση των συστημάτων δημόσιας υγείας και την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές όλων και στις υπονάπτυξη χώρες. Όσον αφορά τώρα τον τρίτο στόχο της χιλιετίας, συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα δράσης για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών. Και για το θέμα αυτό θέλουμε να εμπνευτούμε από τα συμπεράσματα στο οποίο θα καταλήξει το, το Συμβούλιο. Τέλος, θέλουμε να τονίσουμε ότι η Ισπανία σκοπεύει να λάβει υπόψη και τόσα έγιναν στην πρόσφατη διάσκεψη τη Κοπεχάγη και να συνδέσει τις κλιματικές αλλαγές με την ανάπτυξη. Για τους στόχους λοιπόν της χιλιετίας, εμείς πιστεύουμε ότι είναι ο στόχος ο οποίος θα κατευθύνει τις προσπάθειές μας. Δηλαδή, πώς θα πετύχουμε αυτό το στόχο και πώς θα είμαστε αποτελεσματικοί στην αρρωγή μας υπέρ της ανάπτυξης. Η Ισπανία μαζί με την Σουηδική Προεδρία και τις μελλοντικές προεδρίες, την Βέλγικη και την Ουγγρική, θα συνεργαστεί προκειμένου να ετοιμαστεί η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συζήτηση που θα γίνει σε υψηλό επίπεδο στη Σεούλ το 2011 για τους στόχους της χιλιετίας. Πρέπει από τώρα να αρχίσουμε τη δράση μας και γι' αυτό θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στους εξής τομείς. Ε, λογαριασμοί συνεργασία νότου-νότου και καταμερισμός εργασίας. Σε σχέση με το τελευταίο αυτό σημείο και βάσει της δήλωσης της άκρα και με τις εντολές που έχουμε από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεντολογίες για την ε, επικουρικότητα και την καταμονή, κατανομή εργασίας και τα συμπεράσματα του Νοεμβρίου της ΚΑΚΡΗ, η Ισπανική Προεδρία θέλει να βρει πρακτικούς τρόπους για να προχωρήσει το θέμα αυτό της κατανομής εργασίας. Με πρόσφατη μελέτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για τον καταμερισμό, μάλλον τον κατακαιρματισμό ε, της βοήθειας και τις επικαλύψεις που γίνονται πολλές φορές στις προσπάθειές μας, όλα αυτά κοστίζουν πάρα πολλά και αποδυναμώνουν τη βοήθειά μας. Για το κόστος της, ε, του κατακαιρματισμού των δωρητών και της αρρωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας κάνει να χάνουμε κάπου 3 δις 500 ε, εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είμαστε σε περίοδο κρίσης. Είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιες απώλειες όταν είναι περιορισμένοι οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό κυρίες και κύριοι είναι κάτι εντελώς απαράδεκτο και πρέπει να διορθωθεί. Ένας τρίτος παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για τη διάρθρωση της απάντησής μας απέναντι στην κρίση είναι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης και η συνένεση του Monterey που ανανεώθηκε και στην Ντόχα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Ξέρουμε ότι η Ισπανική Προεδρία θα φροντίσει να τηρήσει την εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2009 και να συμπεριλάβει το θέμα των δεσμεύσεών μα όσον αφορά του στόχου τη χιλιετία στη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου. Συγχρόνω θέλουμε το Συμβούλιο αυτό να καταλήξει σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα δέσμευση προκειμένου να πετύχει ο στόχος του 0,7% το 2015. Γιατί έτσι πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη σωστή κατεύθυνση. Επιπλέον, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή μας για τους στόχους της χιλιετίας, πρέπει να υπογραμμίσουμε και την ανάγκη να στηρίξουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να κινητοποιηθούν πόροι υπέρ της δικιάς τους ανάπτυξης. Γι' αυτό θα ήταν καλό να γνωρίζουμε το μέγεθος του προβλήματος. Σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, η ίδια η κυρία Ζολή, μάλιστα, πρόεδρος επιτροπή Επιτροπής αυτής, το δημοσίευσε, λέει ότι για κάθε δολάριο που πηγαίνει στην ανάπτυξη, οι χώρες του Νότου χάνουν 10 δολάρια εξαιτία παράνομων δικτύων. Το συνολικό ποσό των πόρων που χάνονται με αυτόν τον τρόπο είναι κάπου 500.000 μάλλον 500 ε, εκατομμύρια και 800 σε δολάρια κάθε χρόνο. Βέβαια την ευθύνη την έχουν πολλοί. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της προστιθέμενης αξίας που έχει η εμπειρία που διαθέτει σε αυτό το τομέα είναι ένας παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει ώστε να σταματήσει η φοροδιαφυγή. Και γι' αυτό και συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη, ετοιμάζοντας μία ανακοίνωση η οποία να ζητάει ενίσχυση των συστημάτων αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής των υποανάπτυξη χωρών και να προωθήσουμε επίσης ένα διεθνές πλαίσιο συνεργασίας με πρωτοβουλίες όπως είναι το International Tax Compact που πρόθεσε η Γερμανία και που υποστηρίζουμε πλήρως. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι αυτός ο τρόπος εργασίας που έχει να κάνει με τη διεθνή συνεργασία είναι θεμελιώδης. Γιατί όπως είπαμε, οι αιτίε του προβλήματος δεν περιορίζονται μόνο στις υπονάπτυξη χώρες. Πολλές φορές ε, έχω πει ότι η σημερινή, ανέφερα μάλιστα μέχρι τώρα, την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Πρέπει γι' αυτό να δείξουμε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε υπέρ της ανάπτυξης. Καθημερινά να φροντίζουμε για χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Είναι στοιχειώδες να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί χρηματοδότησης που να είναι καινοτόμοι και αυτόνομοι. Ανεξάρτητοι από τη σημερινή συγκαιρία ή από πολιτικές ε, πολιτικά δεδομένα που να βασίζονται στην εθελοντική βάση και στη συνεργασία. Η Ισπανική Προεδρία λοιπόν σκοπεύει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στις εργασίες της ομάδας για την καινοτόμο χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Κυρίες και κύριοι, για τις χώρες ε, ΑΚΕ πρέπει να σας πω ότι ένα από τα κύρια στοιχεία που θέλουμε είναι μια δεύτερη αναθεώρηση της σύμβασης του Κοτονού. Η ενημέρωση αυτή της σύμβασης θα προσαρμόσει τη συμφωνία αυτή σε νέες ε, συμφωνίες σύνδεσης και θα εξυγχρονίσει τις πολιτικές τους σχέσεις, τους θεσμούς τους, τα μέσα και τους μηχανισμούς διαχείρισης ε, που έχουν στη διάθεσή τους υπέρ των στόχων της ηλετίας. και θα ανοίξει η πόρτα σε μη κρατικούς φορείς. Ελπίζουμε αυτό να γίνει καλά και γρήγορα και να υπογραφεί συμφωνία στα πλαίσια τη Υπουργική Συνάντηση Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΚΕ που θα λάβει χώρα στι 3 και 4 Ιουνίου στην Πουργκίνα Φάσο. Στι 27 Μαρτίου μέχρι την 1η Απριλίου στην Τενερίφη από την άλλη μεριά θα γίνει η Ισομερή Συνέλευση Ευρωπαϊκής συνελευση ευρωπαικη ενωση ΑΚΕ. Θέλουμε, όπως και η Προεδρία μας, να προωθήσουμε τη διαδικασία ε, διαπραγματεύσεων προκειμένου να έχουμε νέα μέσα ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν έχει μεγάλη σημασία ε, η εταιρική μας σχέση με την Αφρική, με τη Δυτική Αφρική και ο ΣΕΝΤΕΑ θα παίξει σημαντικό ρόλο για την περιφερειακή ολοκλήρωση. Όσον αφορά την Δυτική Αφρική, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα πολύ καλό πλαίσιο υπέρ της ανάπτυξης της περιοχής με οικονομική και εμπορική ολοκλήρωση. Συνεργαζόμαστε επίσης στενά με τη Βελγική Προεδρία για όλες τις εργασίες που έχουν να κάνουν με την επιτυχία της έσκεψης κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής που θα λάβει χώρα το δεύτερο εξάμεινο του 2010. Θέλουμε όμως επίσης να υποφεληθούμε από την Προεδρία μας για να υπογραμμίσουμε τη σημασία που έχει η συνεργασία της Ευρώπης με την Λατινική Αμερική μέσω της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η νέα κυβέρνηση Ομπάμα έδειξε συμπεριλαμβάνοντα θέματα ανάπτυξης στην ε, ε, διατλαντική ατζέντα ότι δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα. Εμείς Ε, προσκαλέσαμε τον Όριο Σάντα να συμμετάσχει στην Υπουργική Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα λάβει η χώρα στην γράφια στη Σεγκόβια στις 17 και 18 Φεβρουαρίου. Τον Απρίλιο σκοπεύουμε να έχουμε μια πρώτη συνάντηση της συμβουλευτική Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών στη Μαδρίτη. Θέλουμε Μάλλον δεν μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη ένα ηγετικό ρόλο αν δεν στηρίξουμε τους πολίτες μας. Γι' αυτό και σκοπεύουμε να οργανώσουμε διάφορα φόρα και συνεδριάσεις όπου η κοινωνία των πολιτών να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως είπα και στην αρχή, η Προεδρία μας χαρακτηρίζεται από την οικονομική κρίση. Είναι μια στιγμή κατάλληλη για να υιοθετήσουμε μια φιλόδοξη ατζέντα υπέρ της ανάπτυξης και καταπολέμησης των ανισοτήτων και καταπολέμησης της φτώχειας. Πρέπει να μπορούμε να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση δυνατή, ενωμένη για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες των υπονάπτυξη χωρών. Πρέπει να αποφεληθούμε λοιπόν από αυτή την ευκαιρία. Και εμείς θέλουμε με τις πρωτοβουλίες που ανέφερα να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να δείξει την αλληλεγγύη της και να έχει πραγματικές και αποτελεσματικές λύσεις. Υπό την Ισπανική Προεδρία θέλουμε τη δικιά σας στήριξη για να πετύχουν οι στόχοι μας και οι πολιτικοί μας στόχοι να γίνουν πράξη. Είναι πράγματα με τα οποία συμφωνούμε, αλλά και τα οποία μας ενώνουν μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ταυτότητας που έχουμε στον κόσμο. Και το χαρακτηριστικό της ταυτότητας αυτής είναι η αλληλεγγύη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπέρμαν. Δεν φανταζόμουν ότι θα ήσασταν τόσο γρήγορο. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Μωρατίνο. Α, μόνο εγώ σε απογοήτευσα. Ε, φαντάζομαι θα έχει να γνωρίσει και άλλες απογοητεύσει στη ζωή. Σας ευχαριστούμε για την απαρίθμηση των στόχων σας. Ε, Σα συγχαίρουμε ειλικρινά που μέσα τόσο μικρό χρονικό διάστημα προχωρήσατε τόσο πολύ σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ που δίνεται στην αναπτυξιακή βοήθεια. 0,45 ε, από, από 0,40 0,45. Οι άλλες ε, ευρωπαϊκές χώρες πάνε πολύ, είναι πολύ μακριά. Μείωσαν φοβερά το, την αναπτυξιακή του βοήθεια. Η Ιταλία έφτασε στο 0,1%. Σας συγχαίρουμε λοιπόν για, για την προσπάθειά σας και βλέπουμε ότι άλλοι δεν κάνουν ό,τι κάνετε εσείς να επικεντρωθούμε τώρα στην αρχιτεκτονική της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως ε, επαναλαμβάνω πράγματα που έχω ξαναπεί εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Είμαι αναγκασμένος όμως να το κάνω. Γιατί προς το παρόν η Βαρόνη Άστον είναι υπεύθυνη για το μέσο για την αναπτυξιακή συνεργασία. Και ο κ. Πίμπαλξ έχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Δεν υπάρχει συνέπεια εδώ στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση μεταξύ δύο επιτρόπων και μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη της ε, πολιτικής εις βάρος των φτωχών, της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα ήταν πολύ πιο λογικό η κυρία Άστον ε, στο ρόλο της είπα της εκπροσώπου να καθορίσει τις ε, μεγάλες ε, στρατηγικές, ε, τους μεγάλους στρατηγικούς άξονες εποπτείας και ελέγχου και οι δύο μεγάλοι φάκελοι για την ανάπτυξη να είναι υπό την αιγίδα ενός επιτρόπου. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο κ. Μπαρόζο, ίσως γιατί θέλει να είναι έτσι ακριβοδίκαιος με όλους, όλος να πάρει ο καθένα θα πάρει ένα κομμάτι από την πίτα, αλλά δεν είναι λογικό αυτό που έκανε. Δεν είναι... Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πνεύμα τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Δηλαδή, η συνθήκη τη Λισαβόνα λέει να μιλάμε μία φωνή στην εξωτερική πολιτική και, έτσι δεν και όμω δεν πάμε προ αυτή την κατεύθυνση με την κατανομή του κ. Μπαρόζο. Φαντάζομαι, θα ελπίζω τουλάχιστον, η Ισπανική Προεδρία να βοηθήσει, να πείσει για να γίνει μία μικρή αλλαγή προ αυτή την κατεύθυνση που σα ανέφερα. Ο κύριο Μίτσελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήρθα νωρίτερα και καλωσορίζω τον Υπουργό. Ε, το συγχαίρω, δε. Συγχαίρω και την Ισπανία για την πρόοδο που έκανε στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας. Ένα-δύο σχόλια. Τι συζήτηση έχει γίνει πρόσφατα στο Συμβούλιο Υπουργών για να υλοποιηθεί ο στόχος του 0,7%. Η δέσμευση. Όλοι περάσαμε από την κρίση. Και πάντα κατά τη διάρκεια της κρίσης ε, το ΑΕΠ μας συρρυκνώνεται. Άρα και η συνεισφορά μας ε, σε, μειώνεται. Ε, το θέμα είναι να κάνει μια προσπάθεια το Συμβούλιο ε, για να υλοποιήσουμε αυτό, τη δέσμευση του 0,7%. Τι θα κάνει το Συμβούλιο. Ε, τι συζήτηση γίνεται τώρα για τη Χαϊτή. Για την Χαϊτή διάβασα πρόσφατα ότι το 2002 σκοτώθηκαν 2.000 άτομα από έναν σεισμό στην Χιλή, ε, ύψους 9,2 της κλίμακας Ρίχτερ. Τι θα κάνουμε με την ΑΕΤ όμως για να αντιμετωπίσουμε αυτή την καταστροφή. Και τι πιστεύετε για την απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ΑΕΤ. Ήταν συντονισμένη επαρκώς. Υπήρχε ένα αμερικανικό πλοίο το οποίο υποστήριξε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Δεν θα πρέπει και εμείς να έχουμε έτοιμες ε, ομάδες ε, ε, έτσι σε μια κυλιόμενη βάση, ανάλογα με την Προεδρία. Ε, όχι οι Ισπανοί, οι Ιρλανδοί, ο καθένας με την εθνική του σημαία. Δεν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ε, να ανταποκριθούμε σε τέτοιες ανάγκες, τόσο ώστε να παρουσ, ε, παράσχουμε βοήθεια. Δεν θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση για αυτό το θέμα. Δύο γρήγορες ερωτήσεις Κολομβία. Είναι στη μέση διάταξή μας και για τη δολοφονία ε, συνδικαλιστών στην Κολομβία. Ε, υπάρχει πρόοδος στην Κολομβία, αλλά τι έχετε να πείτε για την α, δολοφονία των συνδικαλιστών και πώς θα πιέσετε τον, τον πρόεδρο ούτω ώστε να προστατεύονται τα συνδικάτα. Τελευταίο σχόλιο, κύριε Υπουργέ. Μετά το κόλαφο που λάβαμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κοπενχάγη, όπου οι Αμερικάνοι ξεπέρασαν τους ε, Κινέζους και τους, ε, τους ε, Νοτιοαφρικανούς και έκαναν κάποιες ανακοινώσεις Αλλά τώρα μάθαμε ότι δεν θα έρθει στην ε, σύνοδο του ΟΗΕ ο κ. Ομπάμα. Τι έγινε. Μπορούμε να ρωτήσουμε τι έγινε. Μπορούμε να παίξουμε και σε αυτό το επίπεδο ένα ρόλο. Ε, ξέρουμε ότι σε οικονομικό επίπεδο, όταν ε, το αμερικανικό οικονομικό σύστημα με τα επισφαλή δάνεια ε, κόντευε να καταρρεύσει, παίξαμε το ρόλο μας. Όποτε θέλουν οι Αμερικάνοι Δηλαδή, εμεί κανονίζουμε με βάση το πότε μπορούν οι Αμερικάνοι. Αυτά και σα εύχομαι κάθε επιτυχία ε, για την Προεδρία σα. Η κυρία Σανίκη. Όχι, ο κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Ως Ισπανέος πολίτης, πρέπει να εκφράσω την ικανοποίησή μου και την περηφάνειά μου για τις εξελίξεις στην δικιά μας αναπτυξιακή πολιτική. Ως Ευρωπαίος πολίτης, επίσης πρέπει να στηρίξω τις προσπάθειες της Ισπανικής Προεδρίας προκειμένου ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει φιλόδοξα την αναπτυξιακή της πολιτική. Από αυτήν εδώ την Κοινοβουλευτική Επιτροπή πρέπει να σας πω ότι είμαστε απαιτητικοί και επικριτικοί. Αλλά συγχρόνως είμαστε μια επιτροπή που θα σας στηρίξει πλήρως προκειμένου κατά την περίοδο της Ισπανικής Προεδρίας να επιτευχθούν οι στόχοι που θέλουμε να πετύχουμε όσον αφορά την αναπτυξιακή μας πολιτική. Ορισμένοι από αυτούς ε, αναφέρθηκαν στην αρχική σας παρουσίαση. Και θέλω να αναφερθώ σε έναν από αυτό το στόχο. Ορισμένοι είναι μακροπρόθεσμοι βέβαια, όπως εκείνη του στόχου της χιλιετίας ή όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Άλλοι πάλι ε, ταράζονται κάπως εξαιτίας ε, ανθρωπιστικών κρίσεων ή ηθομηνιών όπως έχουμε στην ΑΕΤ. Τώρα για τους μακροπρόθεσμους στόχους τους στόχους της χιλιετίας, για παράδειγμα. Η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο θέλει το Συμβούλιο να υιοθετήσει ξεκάθαρη θέση το Σεπτέμβριο στη συνάντηση υψηλού επίπεδου του ΟΗΕ για την αναθεώρηση των στόχων αυτών. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει να δραστηριοποιηθεί, αλλά πρέπει συγχρόνως να στηρίξει την επίτευξη των στόχων αυτών. Γιατί οι στόχοι αυτοί δεν μπορεί να μειωθούν ούτε να καθυστερήσουν επειδή είχαμε την οικονομική κρίση από την οποία υποφέρουν οι αναπτυγμένες χώρες. Στηρίζουμε λοιπόν πλήρως την Ισπανική Προεδρία προκειμένου στο Συμβούλιο το Ερινό η Προεδρία να στηρίξει μία δυνατή θέση που να κάνει τη φωνή της Ευρώπης να ακουστεί όσον αφορά την ανάπτυξη και η φωνή αυτή να αποτελέσει παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Έρχομαι τώρα στις κλιματικές αλλαγές. Εδώ είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι. Θέλουμε να στηρίξουμε τις υπονάπτυξη χώρες προκειμένου να προσαρμοστούν ή να τους μεταφέρουμε τεχνολογία, αλλά όλα αυτά μπορεί να αποτελέσουν απειλή για τους πόρους που πάνε στην ανάπτυξη. Εμείς λοιπόν θέλουμε επιπλέον πόρους και όχι να περιορίσουμε τους πόρους που έχουμε υποσχεθεί για την επίσημη αναπτυξιακή αρρωγή. Χαιρόμαστε λοιπόν για τις εργασίες που οδηγούν στην έγκριση νέων πόρων, όπως για παράδειγμα τον φόρο στον οποίο αναφερθήκατε εσείς στην παρουσίασή σας. Τέλος, όσον αφορά την IT, ανησυχούμε ιδιαίτερα. Στο πρώτο στάδιο ανθρωπιστικής αρρωγής πρέπει να υπάρξει και συνέχεια με την ανοικοδόμηση και πάνω απ' όλα να φτιαχτεί ένα κράτος με σταθερότητα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα και δεν φταίει μόνο ο σεισμός. Ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε και επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να βασιστείτε στη στήριξή μας. Όχι μόνο τη δικιά μου που εννοείται, αλλά Είμαι σίγουρος ότι ολόκληρη η Επιτροπή μας θα σας στηρίξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κύριε Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζω με τη σειρά μου τον εξοχότατο προσκεκλημένο μας που παρουσίασε ένα πολύ ε, ενδιαφέρον, πολύ ισχυρό πρόγραμμα σκέπτομαι λίγο τι προσπαθούμε να κάνουμε. Όλοι προσπαθούμε να αυξήσουμε την ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Μιλούμε εδώ για ανθρώπους οι οποίοι ζητούν ε, οι οποίοι ζουν μάλλον με ένα ή δύο δολάρια την ημέρα και θέλουμε να ε, τους φέρουμε σε ένα επίπεδο που να μπορούν να ζουν με τέσσερα ή με έξι. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να επιτύχει η προσπάθεια αυτή όπως είναι. Γιατί και με 6 ευρώ την ημέρα πάλι φτωχή θα είναι. Πρέπει να το εξετάσουμε διαφορετικά. Πρέπει να δούμε πώ οι πλούσιοι πόροι των αναπτυσσόμενων χωρών θα παραμείνουν στι αναπτυσσόμενες χώρες. Που δείχνει και η ε, εκπληκτική μελέτη έρευνα της ε, Εύα Ζολή που έθεσε το θέμα αυτό κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι 500 έως 800 δισεκατομμύρια δολάρια ξεφεύγουν, φεύγουν, εγκαταλείπουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και τα χρήματα που βάζουμε εμείς ξανά, που δίνουμε εμείς στις χώρες αυτές είναι το πολύ το ένα δέκατο. Ναι, μπορούμε να μιλήσουμε για φοροδιαφυγή. Μπορούμε να ε, φτιάξουμε προγράμματα που να επιτρέψουν την επανεπένδυση αυτών των χρημάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου αυτά τα 500-800 δισεκατομμύρια δολάρια να μην εγκαταλείπουν τις χώρες αυτές, να μένουν στις χώρες αυτές και να εργάζονται τα χρήματα αυτά για να αποδίδουν. Τότε θα <clears throat> συμβάλλουμε πραγματικά στην μείωση της φτώχειας. Όπως ο κ. Ντεσότο, ε, πρόεδρος της Βουλής σας, ο οποίο έχει μιλήσει για κινήσεις που γίνονται έξω από τα νομικά πλαίσια, μίλησε για όλες αυτές τις παραγκουπόλεις. που τα όσα παράγονται σε, υπάρχει το κεφάλαιο γιατί είναι ε, ύψος αξίας κάποιων τρισεκατομμύριων δολαρίων. Μπορούμε να τα σκεφτούμε λίγο αυτά. Κύριε Νιούτον, ήταν εσείς. Κύριε Πρόεδρε, μία σύντομη ερώτηση. Ένα από τα μεγάλα ε, συμπτώματα της φτώχειας στην Αφρική είναι και η ροή από ή μέσω της Αφρικής παράνομων ναρκωτικών και παράνομων μεταναστών προς την Ευρώπη. Ποια είναι τα ε, Ποιε είναι οι ιδέες της ε, ισπανική Προεδρίας για την καταπολέμηση αυτών των παράνομων ροών ναρκωτικών και ε, μεταναστών. Ο κ. Γκέρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρω και εγώ την ε, Ισπανική Προεδρία για τι προσπάθειες που αναπτύσσει στην χώρα της και κυρίως για την μείωση του δημοσίου χρέους. Είναι εντυπωσιακέ οι προσπάθειε αυτέ ερώτηση. Δύο ερωτήσεις μάλλον. Πρώτο, τι θα κάνετε με τους διστακτικούς, με τις χώρες εκείνες οι οποίες δεν σέβονται τόσο πολύ τις αρχές ε, της Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την Ανάπτυξη, που προβλέπει να κατέβουμε σε 0,51% το συντομότερο δυνατό και κάτω από αυτό μέχρι το 2015. Άλλωστε έχει γίνει ομόφωνα δεχτεί αυτή η δέσμευση. Δεύτερη ερώτηση, στο ίδιο πλαίσιο, το θέμα που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κοπενχάγη δεν ήταν ιδιαίτερα θετικό και κυρίως για την βοήθεια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του, της του κλίματος για χρήματα τα οποία υποτίθεται θα ήταν πρόσθετα, δηλαδή εκτός της αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτά τα είπαν ορισμένε χώρες, άλλες είπαν ακριβώς, τα αντίθετα. Δηλαδή η Ευρώπη είπε ένα ξεκάθαρο ναι και ένα ξεκάθαρο όχι για το ίδιο θέμα. Δεύτερο, η ορατότητα. Είπατε και σωστά ότι είμαστε ε, οι πρώτοι δανειστές ό,τι αφορά τα ανθρωπιστικά. Τα γνωρίζουμε αυτά εδώ. Έχουμε την εντύπωση ωστόσο ότι εδώ στην Ευρώπη κάνουμε κάθε το δυνατόν για να το κρύψουμε από τον υπόλοιπο κόσμο. Σαν να προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω από μια μαντήλα. μια μπουρκα. Να μην δείξουμε ότι είμαστε οι πρώτοι που δίνουμε πιστώσεις. Δεν πρέπει να το κρύβουμε αυτό από, το, από την κοινή γνώμη. διότι αυτοί που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκονται στο προσκήνιο και η Ευρώπη δεν είναι μεταξύ τους. Τρίτο σύνολο προβλημάτων που θέσατε και σας συγχαίρω η ιδιαίτερη σημασία που δίνεται σε εξωτερικούς παράγοντες που υποθηκεύουν την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κυρίως ύποπτες ε, δημοσιονομικές ε, δραστηριότητες. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί δεν μιλούμε και για τις ε, σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναπτυσσόμενων χωρών, θα δεχθείτε να αναθέσετε μια μελέτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μελετήσει ακριβώς τις επιπτώσεις της αναπτυξιακής βοήθειας από κάθε άποψη και το τρίτο στα πλαίσια της συνοχής των πολιτικών μιλούμε συχνά για τις συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπτυσσόμενων χωρών. Πώς βλέπετε την εξέλιξη της αλληλευτικής συμφωνίας που υποτίθεται ότι θα συναυθεί με το Μαρόκο που εμπίπτει και αυτή στις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής, της ε, Ισπανικής Προεδρίας. Και ποια δυνατό, ποιες δυνατότητες θα δοθούν στου Σαχράουι μέσα στα πλαίσια αυτά. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια που λέτε ότι στηρίζετε τους στόχους της Ισπανικής Προεδρίας. Θα είναι μια πολύ αποτιτική Προεδρία εν μέσω διεθνούς οικονομικής κρίσης, όπως καταλαβαίνετε, αλλά είναι και μια νέα στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε να είμαστε πολίτες του 21ου αιώνα και αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει ένα σημαντικό μήνυμα και να αποτελεί σημείο αναφοράς, πρέπει να δεσμευτούμε υπέρ της αλληλεγγύη και της ανάπτυξης. Κύριε Μπέρμαν, η προσπάθειες της ισπανικής κυβέρνησης δεν είναι 0,48, είμαστε ήδη στο 0,51% για την αναπτυξιακή βοήθεια. Και συνεχίζουμε την προσπάθεια. Το 2008 ήταν 0,48. Ε, Ανεβαίνει. Και την Παρασκευή που μας πέρασε η κυβέρνηση υιοθέτησε μια πολιτική διορθωτική του προπολογισμού με περικοπές σημαντικές, αλλά αποφάσισε η κυβέρνηση να μην αγγίξει ούτε ένα ευρώ από τα όσα είχε αποφασίσει υπέρ της αναπτυξιακής βοήθειας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την απόφαση αυτή της Ισπανικής κυβέρνησης και του Πρόεδρου της. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, ώστε η δέσμευση αυτή, και εδώ απαντάω σε διάφορους που πήραν το λόγο, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο να καταφέρουμε να δεσμεύσουμε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες τις χώρες μέλη προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτός είναι ο στόχος. Μία από τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας όταν ξεκινήσαμε με ή χωρίς Λισαβόνα είπαμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια για πρώτη φορά, για πρώτη φορά, μοναδικό ε, παράδοξο, ποιοι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων κάθισαν και συζήτησαν πολιτικά τη δέσμευσή τους υπέρ της ανάπτυξης. Μετά από 50 χρόνια διαδικασίας ολοκλήρωσης. Τον Ιούνιο λοιπόν 2010 για πρώτη φορά οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων θα κοιταχτούν στα μάτια και θα συζητήσουν και θα πούνε «Ε λοιπόν, τι γίνεται» δεν μπορούμε να δώσουμε 0,51% το 2015 εμείς οι Ευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη μαζί με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να απαλλαγεί από τις ανισότητες και τη φτώχεια. Ε, δεν μπορούμε να κοιταχτούμε στα μάτια τότε αν δεν μπορούμε να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη, αυτή τη δέσμευση. Πρέπει να είμαστε σε θέση. Είμαστε σε έναν ευρωπαϊκό κόσμο που δεν έχει να κάνει μόνο με τους ηγέτες κατών και κυβερνήσεων, έχει να κάνει και με τους πολίτες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι πολίτες θα μας ζητήσουν ευθύνε αν δεν το κάνουμε. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος που θα προσπαθήσουμε να οθήσουμε. Δεν σας εγγυώμαι το αποτέλεσμα, τι θα πούν τα κράτη-μέλη γι' αυτό. Σας εγγυώμαι όμως ότι η Ισπανική Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πετύχει να δεσμευτεί σε αυτό το στόχο. Κύριε Μπέρμεν, με ρωτούσατε επίσης για τη νέα θεσμική αρχιτεκτονική είναι αλήθεια ότι έχουμε μια νέα πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα με μια ύπατο εκπρόσωπο, αντιπρόεδρο της Επιτροπής, με έναν επίτροπο για την ανάπτυξη. Οπότε είναι γνωστό ότι η συνθήκη ε, αναθέτει στην ύπατο εκπρόσωπο ότι έχει να κάνει με την συνεργασία για την ανάπτυξη. Η Βαρόνια Άστον το γνωρίζει πολύ καλά ότι έχει διάφορους χώρους δράσης. Εξωτερική πολιτική, ανάπτυξη, ανθρωπιστική βοήθεια, πράγματα τα οποία μοιράζεται με άλλους επιτρόπους. Βασικό είναι όμως να υπάρχει συνοχή. I want to work on cluster, για να το πω στα αγγλικά, δηλαδή να υπάρχει συνεργασία με άλλους επιτρόπους, διαμορφώνοντας όμως ένα σύνολο πολιτικής. Η Ισπανική Προεδρία θέλει αυτό το νέο στάδιο να διέπεται από συνοχή, να είναι ενιαίο, όπω είπε και ο κύριο Μπέρμαν, και να είμαστε αποτελεσματικοί βέβαια. Ο Επίτροπο για την Ανάπτυξη έχει πολλέ αρμοδιότητε. Αλλά είπα ότι η εκπρόσωπο θέλει να υπάρχει ένα σύνολο για να ενισχυθεί η αναπτυξιακή μας πολιτική. Να είναι ενιαία αντιμετώπιση. Κύριε Μίτσελ, για την ΑΕΤ. Κοιτάξτε λογικά, όταν κάποιος ασκεί την Προεδρία, προσπαθεί να μην αυτοικανοποιείται, αλλά ούτε να είναι και υπερβολικά επικριτικός. Η απάντηση όχι της Ισπανικής Προεδρίας ή της ΥΠΑ της εκπροσώπου ή της Ένωσης, αλλά όλο μαζί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, ήταν εξαίρετη, εξαιρετική, άμεση, γρήγορη, αποτελεσματική. Με μια καταστροφή τέτοιου μεγέθους, το πρώτο που πρέπει να μας απασχολεί, είναι ο κόσμος που υποφέρει οι καταστροφές. Όταν λοιπόν τα Ηνωμένα Έθνη ξεκινάνε με την αρρωγή, την κατεπίγουσα βοήθεια, αμέσως το πρώτο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με την Βαρόνη Άστον πέτυχε 122 εκατομμύρια ευρώ. Αμέσως. που ήταν παραπάνω από το ποσοστό που, ζητούσε, που ζητούσαν τα Ηνωμένα Έθνη. Και παραπάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς. 230 εκατομμύρια ανθρωπιστική βοήθεια. Μετακίνηση μη κυβερνητικών οργανώσεων, εθελοντών. Πέτυχε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια λέει ο Ευρωβουλευτής Μίτσελ ότι η παρουσία της Βόρειας Αμερικής ε, θέτει κάποια ερωτηματικά. Λέει ότι θα θέλαμε μια ευρωπαϊκή δύναμη να φτάνει πριν τους Αμερικανούς. Ε, δύσκολο. Γεωγραφικά, αν μη τι άλλο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, όπω και να το κάνουμε, είναι πιο κοντά στην Αιτία από Η Ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κάνουμε αγώνα δρόμου, ποιο θα φτάσει πρώτο. Κάνουμε αγώνα δρόμου όμω για το συντονισμό και την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Είναι αλήθεια. Με όλες τις κρίσεις, ανα πάσα στιγμή, το μάθημα που πρέπει να παίρνουμε είναι πώς θα βελτιώσουμε τους, οργανισ... τους μηχανισμούς παρέμβασής μας. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Μίτσερ. Δεν επικρίνω αυτά που λέτε, αλλά εξηγώ πώς έχει η κατάσταση. Αλλιώς έχετε δίκιο. Πάντα μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Έτσι λοιπόν και με αυτήν την πρωτοβουλία της Eurofast ή με ανθρωπιστική ευρωπαϊκή δράση που να υπάρχει δυναμικό στρατιωτικό και μη στρατιωτικό, όντως αυτές είναι προτάσεις που θα πάνε στην ΥΠΑ ΕΕ το εκπρόσωπο, ώστε την επόμενη φορά να μπορέσουμε να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Αλλά τα καταφέραμε και το είπαμε αυτό και στην Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη. Υπήρξαν και Ισπανοί και Ιταλοί και Πορτογάλοι και Γάλλοι. Ό,τι θέλετε. Πήγαν και βοήθησαν να γυρίσουν πίσω πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονταν εκεί. Έγινε δουλειά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γρήγορα. Αυτό δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, μπορεί να τα καταφέρει. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να έχουμε ακόμα πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς και θα το φροντίσει αυτό η Πατή Εκπρόσωπος. Μην παραμένουμε όμως στην ανθρωπιστική βοήθεια και την κατεπίγουσα. Όπως είπε και ο κύριος Γερέρο, πρέπει να ξαναχτίσουμε τη χώρα. Μια χώρα σαν την Αιτή που πέρασε από τραγικά γεγονότα και που έτσι κι ήταν μια από τις πιο φτωχές χώρες. Πρέπει λοιπόν να δράξουμε αυτή την ευκαιρία και να αποτελέσει τη δοκιμή, το τεστ, τις εξετάσεις για μας, αν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή. Να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας, όλοι μαζί, και να φροντίσουμε οι δράσεις μας να βγάλουν τη χώρα από αυτήν την μυρολατρεία και να της προσφέρουν ένα μέλλον με ελπίδα. Έρχομαι τώρα στην Κολομβία. Εδώ ξέρω ότι κάποιοι ευρωβουλευτές ανησυχούν με την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κολομβία. Θεμητό. Όλοι πρέπει να ανησυχούμε κάθε φορά που έχουμε συμφωνία με μια χώρα, με μια περιοχή, όπως η συμφωνία με, ανάμεσα στο Σύμφωνο των Άνδεων και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να λαμβάνονται υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας εγγυώμαι ότι και η Ασπανία, η οποία συνεργάζεται με την Κολομβία, εκφράζει ανησυχίες και συνεργάζεται με τις αρχές, τον πρόεδρο Ρίμπερ και άλλους, προκειμένου να καθησυχαστούν οι ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ανοιχτή. Έχουν γίνει συνομιλίες με τις κολομβιανές αρχές και είναι έτοιμοι να ακούσουν προτάσεις. Δείχνουν ότι δεν έχουν καμία δυσκολία να φροντίσουν για μηχανισμούς εποπτείας ελέγχου ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, όπως είπε ο κύριος Μίτσελ, να προστατεύονται στη χώρα αυτή. Τέλος, κύριε Μίτσελ, για την Κοπεχάγη. Κοπεχάγη και αναβολή του, της διάσκεψης κορυφής Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων επίσης τέθηκε αυτό το θέμα σήμερα το πρωί. Οι διατλαντικές ε, σχέσεις βέβαια αποτελούν σημαντικό άξονα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει όλο να το δούμε όμως στο σημερινό πλαίσιο. Είναι περίπλοκη η κατάσταση σήμερα και το γνωρίζετε. Από τις πιο περίπλοκες. Από τη μια έχουν να αντιμετωπίσουμε την ένδια, την απελπισία, την μιζέρια, από την άλλη μεριά κρίση στον κόσμο. Με το θέμα της αναβολής της διάσκεψης αυτής κορυφής δείχνει ότι δεν επήγει το ζήτημα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν νιώθουν ότι επήγει μια τέτοια διάσκεψη. Επήγουν άλλα πράγματα πιο πολύ. Αφγανιστάν, Ιράν. Έχουν δηλαδή διάφορα πράγματα που επήγει να αντιμετωπίσουν, που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια στον κόσμο και οι σχέσεις τους εντάξει είναι με την Ευρώπη. Και πρέπει να βάλουμε περισσότερο περιεχόμενο στις διατλαντικές σχέσεις. Και αυτό θέλει να το κάνει η Ισπανική Προεδρία. Με τις κλιματικές αλλαγές μεταξύ άλλων. Με τον κύριο Φανεροπόη ξέρω ότι συμπεριλαμβάνει ε, στη συνάντηση της 10ης ε, Φεβρουαρίου τη συνέχεια μετά την Κοπεχάγη για να δούμε πώς εμείς οι Ευρωπαίοι μπορούμε να επηρεάσουμε περισσότερο τα πράγματα. Στην Κοπεχάγη αυτό που έγινε είναι ότι δεν ίσχυε η Λισαβόνα ακόμα. Άρα εμείς δεν μπορούσαμε να έχουμε σαφή θέση ενιαία για τις διαπραγματεύσεις. Είχαμε διάφορους διαπραγματευτές. Δεν υπήρχε μία ενιαία ευρωπαϊκή θέση, ένα ενιαίο περιεχόμενο που θα μπορούσαμε να το είχαμε πετύχει αλλιώς για την καταπολέμηση των κλιματικών ε, αλλαγών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ετοιμάσει πολύ καλά τα πράγματα. Αλλά στις διαπραγματεύσεις υπήρξε κάποιος κατακαιρματισμός, γιατί δεν είχαμε τη Λισαβόνα, γιατί δεν υπήρχε ενότητα στην πολιτική μας αντιμετώπιση. Οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων δίχως άλλο θα προσπαθήσουν να το διορθώσουν αυτό, συζητώντας για τη συνέχεια που θα δοθεί στη Κοπεχάγη. Και αυτό θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου. Συμφωνώ με τον Ευρωβουλευτή Γκερέρο από την άλλη για το ότι η συνάντηση αυτή του Συμβουλίου του Ιουνίου προκειμένου να προταθούν και να καθοριστούν οι στόχοι εν ώψη της συνάντησης της Νέας Υόρκης για την αναθεώρηση των στόχων της χιλιετίας, δικό. Είναι αυτή η πολιτική συζήτηση που καλούνται να κάνουν για τις κατών και κυβερνήσεων για να προχωρήσουμε. Οι κλιματικές αλλαγές για τις υποανάπτυξη λοιπόν, χώρες είναι κάτι που απαιτεί να συνεχίσουμε τη βοήθειά μας. Και η Ισπανική Προεδρία λέει επιπλέον πόρους. Υπάρχουν χώρες που λένε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν αυτοί στην αναπτυξιακή βοήθεια. Άλλοι λένε ότι όχι πρέπει να δοθούν επιπλέον πόροι. Διοδείς και την βοήθεια στις υποανάπτυξη λοιπόν, χώρες όσον αφορά την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Κύριε Ντέβα, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Αλλά είναι μια λάθος συζήτηση. Φυσικά, πηγαίνοντας από τα 4 στα 6 ευρώ, σαν team, δεν λύνουμε το θέμα της ανάπτυξης στον κόσμο. Φυσικά και πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για το 0,7%. Η Ισπανική Προεδρία λέει πως ναι, πρέπει. Από την άλλη στην ερώτηση φτάνει, ε, η απάντηση είναι όχι, χρειάζονται και άλλες πολιτικές. Ακριβώς όπως λέει και ο κύριος Δέβα πολύ σωστά, χρειάζονται και άλλες πολιτικές που να επιτρέπουν στις χώρες ε, που αποδέχονται τα χρήματα να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφημιγή, να κάνουν και άλλα πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν αποτελεσματική βοήθεια και με άλλα μέσα, εμπόριο, ανάπτυξη άλλων ευκαιριών στις υποανάπτυξη χώρες. Αλλά το να λέμε ότι το ποσό της επίσημης αναπτυξικής βοήθειας, η προσπάθεια αλληλεγγύης δηλαδή που κάνει η διεθνής κοινότητα, δεν έχει λύσει τις σοβαρές κρίσεις που αντιμετωπίζει η Αφρική, η Λατινική Αμερική, είναι επειδή η επίσημη αυτή πολιτική αργής δεν συνοδεύτηκε από άλλες πολιτικές που να διασφαλίσουν ότι τα χρήματα αυτά πιάνουν τόπο. Συνεπώς, πρέπει να γίνει συμπληρωματική προσπάθεια. Κύριε Νιούτον Ντάν, για τη μετανάστευση. Η Ισπανική Προεδρία Ξέρει, στο Ισπανικό Κοινοβούλιο την κάναμε αυτή τη συζήτηση, τη σχέση μετανάστευση-ανάπτυξη. Αλλά και αυτή είναι μια λάθο συζήτηση, κατά τη γνώμη μου. Γιατί αν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει μετανάστευση. Οπότε, περισσότερη ανάπτυξη για να μην να έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια ροή παράνομων μεταναστών στις χώρες μας. Η Ισπανική κυβέρνηση και η Ισπανική κοινωνία εξεπλάγει. Δεν το ήξερε το πρόβλημα. Το αγνοούσε. Δεν αποτελούσε μέρος της πολιτικής και κοινωνικής της ζωής και δεν λέω ότι το λύσαμε. Η κατάσταση είναι εύθραυστη. Έχουμε όμως αποτελέσματα και σήμερα είμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2007 οι περίφημες σχεδίες, αυτά τα αυτοσχέδια καράβια που φεύγαν από τη Δυτική Αφρική, από την Κάμπια ή από τη Σενεγάλη ή από τη Γουινέα Μπισάο, φτάναν στα Κανάρια νησιά. Πάνω από 5.000 το 2007. Πέρυσι, κανένα. Μηδέν. Γιατί? Γιατί με το Frontex φροντίσαμε να ελέγχουμε και τον ενέριο χώρο, το ότι μας έρχεται από τη Δυτική Αφρική, βοήθησε, βοήθησε. Άρα λοιπόν χρειάζεται ευθύνη από όλες τις πλευρές και με τις χώρες transit. Συζητήσαμε το δράμα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες εκεί. Γιατί βγαίνουν σε τέτοια περιπέτεια, γιατί γίνονται παράνομοι, γιατί δεν κινδυνεύουν τη ζωή τους για να φτάσουν στην Ευρώπη. Και αναπτύξαμε κάποιες πολιτικές συνεργασίες με αυτές τις χώρες, προκειμένου οι χώρες αυτές να μπορέσουν να ε, βοηθήσουν ε, στη γεωργία, στην κατάρτιση, την ανάπτυξη γενικά. Τις βοηθήσαμε τις χώρες αυτά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια δεν χρειάζεται, χρειάζονται και άλλες πολιτικές, στις χώρες προέλευσης μεταναστών. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζονται συνοδευτικά μέτρα και εκπόνηση σφαιρικών πολιτικών ανάπτυξης. Θα φέρουν αποτελέσματα. Θα περιορίσουν την μεταναστευτική πίεση. Θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, απατώντας και στον κύριο Κόρης για το 07, είπα ότι είναι ο στόχος που θα προτείνουμε στο Συμβούλιο. Και πρέπει να πολεμήσουμε γι' αυτόν. Τώρα, τι προβολή έχουμε. Και χτες το έλεγα στο Γενικό Γραμματέα όταν ετοίμαζε αυτή τη συνάντηση. Βυρμανία, για παράδειγμα, Κίνα. 130 εκατομμύρια δίνει η Κίνα. Μόνη της, ε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Πάνω από 150. Ναι. Είναι ορατή η βοήθεια αυτή εκεί. Οι αρχέ η Βερμανία θεωρεί την Κίνα συνομιλητή τη. Δεν θεωρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν καταλαβαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη δίνει τα 155 εκατομμύρια. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο διαθέτουμε πόρους. Έχουμε μία μελέτη αυτή την εποχή για τη συνολική αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρικανική Ήπειρο. Χρειάζεται. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αν έχουμε αποτελέσματα. Είμαστε οι πρώτοι δωρητές στην Αφρική. Την Κυριακή που μας ε, πέρασε, συνάντησα τον πρώτο Σαδίσα Βέμπα και συζητούσαμε για την Αφρικανική Ήπειρο. Εμάς τους Ευρωπαίους μας κοιτούν με ενδιαφέρον, αλλά από απόσταση. Μας βλέπουν μακρινούς. Πολλοί Αφρικανοί ηγέτες λένε ότι η Ευρώπη το μόνο που θέλει είναι να έχει κάποια υποπτία στην Αφρική, αλλά όχι να μας βοηθήσει πραγματικά. Εμείς τους βοηθάμε να μην πεθάνουν, ως εκεί, τίποτα παραπάνω. Δεν βοηθάμε να αλλάξει η Αφρικανική Ήπειρος. Αυτό δεν έχει γίνει. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με πολιτικές αναπτυξιακές συνεργασίες διαφορετικές, σφαιρικές, που να συμπεριλαμβάνουν όλες, τη... όλες τις χώρες μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί. Αυτό θα μας κάνει περισσότερο ορατούς. Όχι το να σηκώνουμε τη σημαία μας και να φαίνεται η σημαία μας, όπως είπαν μερικοί, γιατί είπαν να δεν υπήρχε η ευρωπαϊκή σημαία στην ΑΕΤ, δεν την έβλεπε κανείς. Μα δεν είναι αυτό. Είναι γιατί η δράση δεν είναι αρκετά αποτελεσματική. Πρέπει να αλλάξει η πραγματικότητα επιτόπου με τη βοήθειά μας. Και τότε όλοι θα ξέρουν ότι η αλληλεγγύη που επέδειξε η Ευρώπη ήταν το καθοριστικό για να αλλάξει η κατάστασή τους. Τέλος, όσον αφορά τις αλληλευτικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μαρόκο είναι ένα θέμα που θα εξετάσει η Επιτροπή Αλίας. Και εγώ έχω εμπιστοσύνη στις αρμοδιότητες των επιτροπών σας, οπότε δεν θέλω να αναμειχθώ σε αυτό το θέμα. Ε, μόνο θα πω ότι υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Πρέπει φυσικά να περιμένουμε τη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποφανθεί επ' αυτού. Η Ισπανική Προεδρία έχει τη νομική υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών που επέτρεψε την εκμετάλλευση της συμβάσης με διάφορους διεθνείς φορείς και αναγνώρισε την ε, δίκηση του Μαρόκο στη Δυτική Σαχάρα. Τώρα από εκεί και πέρα τα κέρδη, τα ωφέλη πρέπει να πάνε στον λαό της Δυτικής Σαχάρας. Τώρα δεν θα έλα να μπω εδώ σε συζήτηση για το τι έδωσε η μαροκινή κυβέρνηση εκεί και τι όχι. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι είναι περισσότερα από πλευρά επενδύσεων. Αλλά αυτή είναι μια πολιτική συζήτηση. Δεν νομίζω ότι είναι εδώ ο πιο κατάλληλος χώρος. Πάντως, το σημαντικό που πρέπει όλοι να στηρίξουμε είναι να βρεθεί οριστική και πραγματική λύση στο πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας. Έχουμε καλά νέα. Από ό,τι φαίνεται θα ξαναρχίσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στο Μαρόκο και το Πολυσάριο, το μέτωπο Πολυσάριο. Δεν νομίζω ότι ξέχασα τίποτα κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν και άλλοι βουλευτέ που θέλουν να πάρουν το λόγο. Κυρία Ζήμερ. Εκφράζω τον σεβασμό μου για τον ενθουσιασμό που επιδείξατε και μακάρι και μερικοί υπουργοί ανάπτυξης κάποιων ευρωπαϊκών χωρών μελών, μακάρι να είχαν και αυτοί, οι οποίοι δεν έχουν άλλο χαρτοφυλάκιο, μόνο αυτό έχουν τη ανάπτυξη, να δείχνουν τέτοιο ενθουσιασμό. Σε πολλές από τις θέσεις που αναφέρατε και ως στόχους, τις συμμερίζομαι απόλυτα. Θα πω τώρα, θα αναφερθώ σε τρία πράγματα. Αφενός Κοπενχάγη και τα αποτελέσματά της, τα οποία ήταν απογοητευτικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες, πολλοί από τους εταίρους μας, αναπτυσσόμενες χώρες και δεν εννοώ μόνο τους κυβερνητικούς εκπροσώπους αλλά και τα NGO, επέκριναν όχι μόνο τα ανεπαρκή αποτελέσματα της ε, Κοπενχάγης αλλά και την έλλειψη προθυμίας μέχρι τώρα να αναλυθεί αγώνας κατά των ζημιών, των βλαβών που προκαλεί η αλλαγή του κλίματος και ιδίως στις πιο φτωχές χώρες. Γιατί αυτές οι πιο φτωχές χώρες είναι αυτές που πλήττονται και περισσότερο από τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος. Και πάλι μέσα σε αυτές τις φτωχές χώρες πάλι τα φτωχότερα στρώματα, αυτά που ζουν δηλαδή με ένα άπειρο ελάχιστο εισόδημα. Εδώ πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικοί στόχοι και να αναπτυχθεί μια νέα νοοτροπία. Δεύτερο, στην ακρόαση των υποψηφίων επιτρόπων, πολλοί αναφέρθηκαν στην αυστηρή διάκριση μεταξύ σταθιωτικών παρεμβάσεων και αναπτυξιακής βοήθειας που χορηγείται και με τη βοήθεια NGO και ζήτησαν να υπάρχει σαφής, ξεκάθαρη διάκριση κυρίως από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από πλευρά χώρων μελών. Πώς το βλέπετε εσεί, θα ζητήσετε από το Συμβούλιο γιατί υπάρχουν και υπουργοί οι οποίοι για να χορηγήσουν αναπτυξιακή βοήθεια, για παράδειγμα στο Αφγανιστάν, θέλω ένα παράδειγμα τώρα, απαιτούν η χώρα να δεχθεί και στρατιωτική παρέμβαση θα το θέσετε αυτό στο, στα πλαίσια του Συμβουλίου Υπουργών Ανάπτυξης για να πείτε ξεκάθαρα και να επιμείνετε ότι δεν επιτρέπεται να τεθούν σε κίνδυνο πρωτοβουλίες χορήγης ανθρωπιστικής βοήθειας με τέτοιες απαράδεκτες απαιτήσει όπως της δεκτυρικής παρέμβασης. Και επίσης Μιλήσατε αρκετά εκτεταμένα και για τον προβληματισμό με τους παράνομους μετανάστες και στην Ισπανία και για τη στρατηγική που προτίθεστε να ακολουθήσετε. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα. Λέτε ότι η χρήση του καθεστώτος Frontex οδήγησε κυρίως ότι δεν μπόρεσαν πλέον να προσεγγίσουν τα Κανάρια νησιά άλλα μικρά σκάφη προτίθεστε να κάνετε παρόμοια πράγματα και για τη Μάλτα, την Λαμπεδούσα στην Ιταλία. Συμφωνώ με αυτά που λέτε στη στο δεύτερο μέρος της απάντησής σας για την χορήγηση περαιτέρω αναπτυξιακής βοήθειας στις χώρες όπου προχωρούν οι μετανάστες. Αλλά για το πρώτο θέλω πιο πολλές λεπτομέρειες. Δεν προέβλεπα να μιλήσω, αλλά χαίρομαι που έχω την ευκαιρία. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, το πρόγραμμά σας είναι πολύ φιλόδοξο και πολύ σημαντικό και είμαι πεπισμένη ότι η Ισπανία κυβέρνησή της θα κάνει θαυμάσια δουλειά. Μιλήσαμε για την ΑΕΤ. Είναι σαφές ότι η προτεραιότητα των, της βοήθειας πηγαίνει σε αυτή την καημένη χώρα. Εγώ πρόσφατα επισκέφθηκα και την Αγγόλα. Είναι μια χώρα η οποία δηλώνει ότι παπάει μια χαρά στην Αφρική, δεδομένη της καταστροφικής κατάστασης της Αφρικής. Τώρα, θα ήθελα να επανέλθω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στους λαθομετανάστες. Είναι ένα σοβαρό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ιταλία. Θα πρέπει να ασχοληθεί και να επιφορτιστεί και η Ευρώπη με αυτό το θέμα. Και θα πρέπει να θέσετε εσείς, κύριε Υπουργέ, αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν ε, πλοία, βάρκες δηλαδή, ε, οι οποίοι, ξέρετε, δεν πηγαίνουν προς την Ισπανία. Όλα τα, τα σκάφη αυτά φτάνουν στην Ιταλία. Ε, αυτό το βάρο το φέρουμε μόνοι μας. Θα πρέπει κάποια στιγμή και η Ευρώπη να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κυρία Στρίφλερ. Προηγουμένως είπατε ότι το να εφαρμόσω μια διαφορετική πολιτική, ότι να γίνουν ορατές οι επιπτώσεις της αναπτυξιακής πολιτικής. Συμφωνώ να το κάνουμε. Επίσης είπατε, σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, ε, το, το, το θέμα δεν είναι να φαίνεται ότι δίνουμε ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά να είναι αποτελεσματική. Είναι ανθρώπινο κάθε ηθήνων οποιασδήποτε χώρα να θέλει να δείχνει τι έκανε η χώρα του. Αλλά οι πολίτε τη δική μου χώρα ποτέ δεν με ρωτάνε τι έκανε η Γαλλία. Με ρωτάνε τι κάνει η Ευρώπη. Και πραγματικά αισθανόμαι κάπω αμήχανα να του απαντήσω. Εντάξει, του είπα τι έκανε η Ευρώπη, αλλά δεν είναι γνωστό τι κάνει η Ευρώπη τελικά. Θα ήθελα να επιμείνω για τη σημασία, όπως είπε ο κ. Μίτσο, να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό φορέα, αν θέλετε. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να γνωρίζουν τι κάνει η Ευρώπη με τα κονδύλια που έχει στη διάθεση, με τα κονδύλια τους, με τα κονδύλια των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Δεν νομίζετε ότι υποτιμάτε λιγάκι την ε, ορατότητα αυτή και ότι ο πολίτης όχι μόνο έχει δικαίωμα να ξέρει, όχι μόνο το, την, την υποχρέωση, αλλά και το δικαίωμα να ξέρει. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια, κύριε Υπουργέ, για τα σχέδια και το πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας. Και εγώ ε, ενθουσιάζομαι με το ενθουσιασμό σας και το πάθος της Ισπανίας οφείλεται στην ιστορία της, οφείλεται και στην πρόσφατη ιστορία της. Ε, δεν θα κάνω μακρές δηλώσεις, ε, θα το ακούσετε αυτό με χαρά, αλλά θα ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε ή διαφωνούμε, διαφωνείτε ότι μπορούμε να ασχοληθούμε με τη λαθομετανάστευση από την Αφρική όταν εξαλειφθεί ο πόλεμος, ε, η απελπισία και τα βασανιστήρια. Όλα τα είναι εμβαλωματικές λύσεις, συμφωνείτε θα πρέπει να, όντως να κάνουμε πρόοδο προς τους στόχους της χιλιετίας. Εσείς ως Προεδρία ε, ετοιμάζεστε για την θέση της Ευρώπης ε, στη Σύνοδο Κορυφής το Σεπτέμβριο ε, για τους στόχους της χιλιετίας συν 10. Τώρα, τι θα κάνει η Ισπανική Προεδρία ούτω ώστε να επανευθυγραμμίσουμε του στόχου τη χιλιετία και να θέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο στην καρδιά αυτής τη πρωτοβουλία, αλλά στην πρωτοβουλία για την επανέναρξη ενό ε, παγκόσμιου διαλόγου για την αποτελεσματική ανάπτυξη. Αυτέ οι δύο ερωτήσει, παρακαλώ. Και τώρα ας πάρω και εγώ το λόγο. Πραγματικά αισθάνεται κανείς καλά όταν ακούει τόσο ενθουσιώδεις ομιλητές ε, και όταν ε, ο ενθουσιασμός αυτός είναι από την Προεδρία του Συμβουλίου και μάλιστα όταν ακούμε και οικονομικές δεσμεύσει από αυτό το κράτος μέλος. Και χαίρομαι που επιτέλους τα θέματα της ανάπτυξης είναι γεγραμμένα στην ατζέντα του Συμβουλίου κατά προτεραιότητα. Θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήματα. Λέτε ότι η κυρία Άστον θα ε, συνεργαστεί με τους υπόλοιπους επιτρόπους ε, και ότι πραγματικά ενδιαφέρεται τα μάλλα για την αναπτυξιακή πολιτική. Πώς εξηγείτε τότε που στο ιδιαίτερο γραφείο της δεν έχει ούτε έναν ειδικό για αναπτυξιακά θέματα, ούτω ώστε να εξασφαλίσει το σύνολο των εξωτερικών πολιτικών συντονίζονται σωστά και λαμβάνουν υπόψη την αναπτυξιακή διάσταση. Αυτό με ανησυχεί, αυτή η έλλειψη. Και δεύτερον, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας για την για τον ακριβή καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ της κυρίας Άστον, του κυρίου Πίμπαλξ και των υπολείπων επιτρόπων αρμοδίων. και την Επίτροπο για την Ανάπτυξη. Έπειτα, Είσαστε ήσασταν αποτελεσματικοί ε, στη βοήθεια που χορηγήσατε στην IT, ε, χάρη στο γεγονός ότι είχατε ήδη επιτόπου ε, ομάδες στον Παναμά, κοντά δηλαδή. Δεν θα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοια διευθέτηση έτσι, σε μόνιμη κατάσταση, να έχουμε τέτοιες ομάδες. Ο κ. Μπέρμαν, μία ενημερωτική ερώτηση. Ο κ. Ντίβα έκανε ε, υπολογισμό. Δεν είναι 4 ή 6 σεντ, είναι 40 ή 50. Αν διαιρέσει το ποσό με τους ανθρώπους. Και το... Και τον προϋπολογισμό 71,3 ευρώ. Επομένως, όχι 4 ή 6 σεντ, αλλά 50. Ο κύριος Ασένης, συντομότατα παρακαλώ. Λύσαμε, μιλήσαμε για την μετανάστευση. Πολύ. Μέχρι το 2050 λέμε ότι οι πρόσφυγες θα γίνουν 500.000. Σήμερα είναι 20.000. Εκατομμύρια, συγγνώμη. Στη Ρουάντα, στην Αιθιοπία, έχουμε διάφορα προβλήματα με τα δάση. Άρα η παραγωγή γεωργική μειώνεται, ε, το νερό μειώνεται, ε, αλλά έχουμε προγράμματα για να προσαρμόσουμε, ε, για να κάνουμε κάποιες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη νερού. Εσείς θα γνωρίζετε αυτά τα προγράμματα, είσαστε διατεθειμένος να βοηθήσετε να προωθήσετε αυτές τις πρωτοβουλίες, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίζει περισσότερο αυτά τα προγράμματα έτσι, α, μείωσης της φτώχειας και της ένδυας. Ε, κύριε Υπουργέ, έχετε 10 λεπτά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Ήδη σας κάνουν υπερορίες τώρα οι διερμηνείς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ελπίζω να μην ξεχάσω καμία ερώτηση. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Για την Κοπεχάγη πάλι. Είναι αλήθεια ότι όλοι απογοητευτήκαμε γιατί είχαμε βάλει στοίχημα όλοι οι Ευρωπαίοι να πετύχουμε μια δεσμευτική συμφωνία στην Κοπεχάγη. Όμως δεν τα καταφέραμε. Η Ευρωβουλευτής που το υπενθύμησε, έχει δίκιο ότι αυτοί που πλήττονται κυρίως από τις κλιματικές αλλαγές δεν είμαστε οι πολίτες του αναπτυγμένου κόσμου, αλλά οι χώρες που υποφέρουν από ένδια και από χαμηλότερα επίπεδα ανάπτυξης. Εκείνοι πλήττονται περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως με περηφάνεια μπορούμε να πούμε ότι γι' αυτό και έχουμε ένα ταμείο για την προσαρμογή όλων των χωρών και η ισπανική θέση είναι σαφής ότι χρειάζονται επιπλέον πόροι και δεν πρέπει να αφαιρέσουμε πόρους από την γενική αναπτυξιακή αρρωγή. Η δεύτερη ερώτηση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι η διαλεκτική αυτή που υπάρχει. Από τη μια συνεργασία και στρατιωτική Όλοι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια. Πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα νοοτροπία συνεργασίας. Υπενθυμίσαμε την εμπειρία από το Αφγανιστάν. Μπορώ να σας πω ότι η πρώτη προσπάθεια του Υπουργείου Συνεργασίας και Ανάπτυξης να βοηθήσει για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στο Αφγανιστάν άκουσε πολλές αντιρρήσεις και υπήρξε και απόρριψη. Απόλυτη οι άνθρωποι που δουλεύουν για τη συνεργασία να μπουν υπό, μάλλον όχι, υπέ, ούτε καν, υπό, ούτε καν να συνεργαστούν με τους στρατιωτικούς δεν θέλανε. Γιατί ήταν δύο διαφορετικές νοοτροπίες που αντιτίθενται μεταξύ τους. Όταν βλέπει κανείς ένα στρατιωτικό, αμέσως σκέφτεται ότι την αλληλεγγύη την απορρίπτει ο στρατιωτικός. Αυτό όμω αρχίζει να αλλάζει αυτή η νοοτροπία. Δεν είναι εύκολο, αλλά για παράδειγμα αυτή η προσπάθεια που κάνουμε για αλλαγή στην νοοτροπία όσον αφορά την συνεργασία, την ανάπτυξη και το στρατιωτικό τομέα, στο Αφγανιστάν, εκεί που είναι παρούσα η Ισπανία, πρέπει να σας πω ότι εκεί υπάρχει αλλαγή. Υπάρχει συνεννόηση πια και κατανόηση και από τις δύο πλευρές για το τι μπορεί να προσφέρει κάθε πλευρά. Είναι δύσκολη η συνεργασία και η ανάπτυξη του Αφγανιστάν αν δεν υπάρχει ασφάλεια. Και δεν υπάρχει ασφάλεια αν δεν υπάρχει ανάπτυξη. Άρα λοιπόν το να μιλάμε απομονωμένα ο ένας από τον άλλον δεν έχει νόημα. Και τα δύο πρέπει να μπουν μαζί. Όλοι να κάνουμε προσπάθεια για καλύτερη αμοιβαία κατανόηση. Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις όταν λοιπόν. πήγαν οι στρατιώτες από τη Βόρεια Αμερική στην Αιτή. Ε, υποθέτω ότι ο κόσμος που ασχολείται με την ανάπτυξη έφρυξε. Αμάν, μόλυνση, ρήπανση, εντός αγωγικών βέβαια. Η προσπάθεια αλληλεγγύης ρηπαίνεται εντός αγωγικών πάντα από τη στρατιωτική παρουσία. Δεν είναι αλήθεια όμως. Δεν είναι αλήθεια. Γιατί και αυτοί βοηθούν για την αλληλεγγύη, αλλά υπάρχουν τέτοια κλισέ που εμένουν στα μυαλά των ανθρώπων δυστυχώς. Όλοι λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια. Οι στρατιωτικές δυνάμεις πρέπει να στραφούν και να δουν διαφορετικά την τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι οποίε με τη σειρά του πρέπει να στραφούν προ τι στρατιωτικέ δυνάμει και να αντιληφθούν ότι έχουν άλλη αποστολή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε τις δομές εκείνες που θα βοηθήσουν δυνάμεις και του στρατού και των μη κυβερνητικών οργανώσεων να πάνε εκεί που μπορούν να προσφέρουν το καλύτερο και ο καθένας να έχει το δικό του ρόλο. Αλλά η σύλληψη είναι σφαιρική υπέρ της συνεργασίας και της ανάπτυξης. Για τη μετανάστευση τώρα δεν θέλω να επανέλθω, γιατί Frontex είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Φέρει σε πέρας μια πολύ καλή αποστολή και προστατεύει τα σύνορα πράγμα το οποίο δεν το αντιλαμβανόμαστε πάντα σε όλο του το μέγεθος, χάρη στη Frontex σώθηκαν πάρα πολλές ζωές. Γιατί από αέρος ή στη θάλασσα η Frontex βρίσκει ναυάγια ή τέλο πάντων βάρκες, σχεδίες που κινδυνεύουν να καταλήξουν σε ναυάγιο και αυτή ακριβώς η εποπτεία είναι που βοηθάει να σωθούν πολλές ανθρώπινες ζωές. Και μετά ακολουθούν βέβαια την διαδρομή επαναπατρισμού εφόσον πρόκειται για παράνομους. Η Frontex λοιπόν είναι αναγκαία και πρέπει να αναπτυχθεί με, με περισσότερους μηχανισμούς, όχι κατασταλτικούς, εποπτείας, προστασίας, διασφάλισης των συνόρων μας. Δεν φτάνει η Frontex οι ροές αυτές παράνομης μετανάστευσης για να αντιμετωπιστούν χρειάζεται περισσότερη συνεργασία, περισσότερη σταθερότητα, περισσότερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελπίδα στην Αφρικανική Ήπειρο. Για την κυρία Σανίκη, έχετε δίκιο σε έναν βαθμό. Η κατάσταση στην Ισπανία όντω έχει βελτιωθεί. Αλλού στην Ευρώπη είχαμε δύσκολες στιγμές τώρα για τις σχέσεις της Ιταλίας με Λιβύη λύθηκε κατέρωθεν ευθύνη και βελτιώνεται και εκεί κάπως η κατάσταση. Όμως είναι αλήθεια ότι το παράνομο κύκλωμα, οι μαφίες κινητοποιούνται και στην Ισπανία. Ξεκίνησαν στα σύνορα με το Μαρόκο, στο Θέουτα και στη Μαλίγια, να δραστηριοποιούνται. Όταν έχουμε μια καλή συμφωνία με το Μαρόκο, Μα ερχόντουσαν από την Μαυριτανία οι μετανάστες. Όταν είχαμε μια καλή συμφωνία με την Μαυριτανία ερχόντουσαν από την ε, Γουινέα Βισάο και όταν είχαμε μια καλή συμφωνία με αυτή τη χώρα από τη Σενεγάλη και ούτω καθεξής. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια σφαιρική αντιμετώπιση όχι μόνο για την ε, Δυτική Αφρική, ή για τη Βόρεια Αφρική ή να μιλάμε για την ε, Μεσόγειο, την Ελλάδα, την Κύπρο, τα λίγα κτλ. Χρειάζεται μια σφαιρική αντιμετώπιση ώστε οι ροές Παράνομη μετανάστευση, είτε μας έρχονται από την Ασία, είτε από το κέρας της Αφρικής, την Ερυθρέα, τη Σομαλία. Γιατί μας έρχονται. Γιατί υπάρχει αστάθεια στις χώρες τους. Άρα λοιπόν πρώτα πρέπει να λυθούν οι ρίζες του προβλήματος και μετά να μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε αποτελέσματα. Αφρική, ναι, έχουμε πάρα πολλέ μεγάλες χώρες με οικονομικές δυνατότητες και άλλες όχι, με τεράστιες δυσκολίες οικονομικές. Γι' αυτό πρέπει με την εξωτερική μας δράση να φροντίζουμε και την Αφρική. Στην κυρία Σουφλέρη για την ορατότητα, ε, για την προβολή που έχει η Ευρώπη και την αποτελεσματικότητά της. Φυσικά και χρειάζεται να υπάρχει κάποια προβολή, ναι. Τι κάνουμε Ευρωπαίοι. Δεν μας βλέπουν, δεν μας βλέπει ο κόσμος, δεν προβάλλουμε τη δράση μας. Γιατί, γιατί δεν αξιοποιούμε αυτό που κάνουμε. Είμαστε συνέχεια επικριτικοί απέναντι στους αυτούς μας, ενώ το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αξιοποιούμε τη δράση μας. Να την λέμε, να την φωνάζουμε. Πρέπει να το πούμε στους Γάλλους ότι είναι όλα η Ευρώπη. Αν λέμε ότι η βοήθεια πήγε αμέσω, ότι είχαμε 500 μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δραστηριοποιήθηκαν για να σώσουν ανθρώπινες ζωές, ότι στείλαμε πάνω από 150 αεροπλάνα, αν τα λέμε αυτά στη γαλλική κοινή γνώμη θα το μάθει. Αλλά αντί να κάνουμε αυτό, τι κάνουμε. Λέμε, α, οι άλλοι τα έχουν καταφέρει καλύτερα από μας. Μα είναι σαν τρεπόμαστε για αυτά που κάνουμε. Να αναγνωρίσουμε ότι προχωράμε, ότι προδεύουμε. Λοιπόν, πρέπει να νιώθουμε περήφανοι για τα καλά που κάνουμε και να το λέμε και να το φωνάζουμε. Δεν λέω ότι δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καλύτερο συντονισμό της δράσης μας, ναι. Ο Ευρωπαίος πολίτης αυτό θέλει να ξέρει. Τι κάνει η Ευρώπη. Και πρέπει να έχει την ικανοποίηση για τα λίγα και καλά που κάνει η Ευρώπη. Κύριε Κάσμαν για το τι κάνει η Ισπανική Προεδρία. Κοιτάξτε, η διάσκεψη της Νέας Υόρκης θέλουμε να στεφθεί από επιτυχία. Πρώτα απ' όλα, θα φροντίσουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επιβεβαιώσει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Πρέπει από τους 8 στόχους για τον καθένα να δούμε πώς εξελίχθηκε. Άλλος προχώρησε περισσότερο, άλλος λιγότερο, να κάνουμε τη διάγνωση. Πού βρισκόμαστε, τι καθυστερήσεις υπάρχουν για τον κάθε ένα από αυτούς τους 8 στόχους. Μπορεί να έχουμε βέβαια την τάση να επικεντρωθούμε σε έναν ή σε δύο. Δεν πρέπει όμως, πρέπει να εξετάσουμε όλους τους στόχους, πώς έχουν προχωρήσει. Και μετά το βασικό, να φροντίσουμε για την βιωσιμότητα να αντέξει η προσπάθεια αυτή, η στήριξη αυτή να συνεχιστεί. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να φροντίσουμε η ευρωπαϊκή προσπάθεια υπέρ των στόχων της χιλιετίας να συνοδευτεί από αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση. Θα δουλέψουμε λοιπόν γι' αυτό για να ενισχυθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κυρία Ζολή, την πρόεδρο. Κυρία Πρόεδρε, ξέρω ότι οι προσδοκίες είναι πολλές, ανυπομονησία επικρατεί. Όχι μόνο στις επιτροπές, αλλά και στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, στα μέσα ενημέρωσης. Πώς προχωράει η νέα συνθήκη της Λισαβόνας, πώς εφαρμόζεται τα νέα θεσμικά όργανα ή πώς προχωράμε, πώς δουλεύουμε. Υπάρχει ανυπομονησία. Α είμαστε όμω λίγο υπομονητικοί. Ένα μήνας μόνο έχει περάσει. Και η Βαρόνη Άστον φτιάχνει την ομάδα με τους συνεργάτες της. Συνδυάζουμε γραμματεία του Συμβουλίου, Επιτροπή. Αυτά είναι πράγματα που θέλουν δουλειά. Εγώ ξέρω τη δικιά μου εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας αφήσουμε το χρόνο να δουλέψει. Η Βαρόνη αναμφίβολα θα έχει κάποιον στην ομάδα της που θα μπορέσει να παρακολουθήσει τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Ακόμα όμως δεν τους έχει φτιάξει τους συνεργάτες της, δεν τους έχει ε, βάλει στις θέσεις τους. Πρώτα οργανώνει τους συνεργάτες της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει τη θητεία της. Άρα λοιπόν δεν έχουμε αρχίσει καλά-καλά. Και μετά θα δούμε το ρόλο των επιτρόπων, τη σχέση μεταξύ τους. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από την κατανομή όταν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων έχει ξεκινήσει, τότε θα δούμε τι πρόγραμμα έχει, τι σχέσεις θα έχει με τους υπόλοιπους και τότε θα ξέρουμε τι κάνει ακριβώς ο καθένας.